Να αρχίσουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Πάμε στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας στο Brexit. Θα συζητήσουμε βάσει του σχεδίου μελέτης ε, για τις πιθανές επιπτώσεις του Brexit πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως ε, γνωρίζουμε, η Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι θα δρομολογήσει το άρθρο 50 ε, στις 29 Μαρτίου για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κρίμα για μας. Θεωρώ ότι είναι θλιβερό αυτό, ειδικά που σήμερα έχουμε και την 60η επέτειο από τη Συνθήκη της Ρώμης. Δεν μπορώ να κρύψω την απογοήτευσή μου. Ε, αλλά αυτό αποφάσισε το Ηνωμένο Βασίλειο, την έξοδο από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητήσαμε με τους συντονιστές τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μελετήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις. Ε, δώσαμε μάλιστα και υλικό ε, στον Κίφερ Χόφστατ για την συζήτησή του με τον Μισελ Μπαρνιέ Είχαμε πει όμως ότι θα το συζητήσουμε και εντός της Επιτροπής μας αυτές τις πιθανές επιπτώσεις και για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τη δουλειά μας, η Επιτροπή μας ε, έχει ορίσει τον Σαλ Γκέρνς ε, για την, Gerns, για την ε, συντονιστή για την συζήτηση αυτή που αφορά τις τις επιπτώσεις του Brexit πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα επόμενα χρόνια. Οπότε, ε, εκτός από τον κύριο Γκέρενς, χρειαστήκαμε και κάποια βοήθεια εμπειρογνωμόνων εξωτερική. Ελπίζω να έχετε μία, ένα αντίτυπο της μελέτης. Φαντάζομαι την έχετε στη διάθεσή σας. αν υπάρχουν ε, αντίτυπα μπορούμε να τα διανύμουμε και σε όσους δεν τα έχουν, αλλιώς ε, υπάρχει και στον ιστότοπο η μελέτη. Πάντω αν υπάρχουν αντίτυπα επιπλέον μπορεί να ρίξουν μια ματιά όσοι ενδιαφέρονται. Η Λιάννα Ολιβιέ που είναι ανώτερη αναλύστρια και, αναλύτρια και Αίτορ Πέρες ε, από το, Ελκάνο, το Ινστιτούτο Ελκάνο στην Μαδρίτη. Έκανα λοιπόν μια μελέτη για το τι θα μπορούσε να συμβεί, ποια είναι τα ζητήματα που αφορούν το Brexit και χαίρομαι όλους ιδιαίτερους που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι η αρχή, η διαδικασία, η αρχή της διαδικασίας και του προβληματισμού μας. Με πολύ χαρά θα ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Δεν ξέρω από ποιον θέλετε να αρχίσουμε. Κυρία Ολιβιέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα. ομιλήτρια. aunque, el informe está redactado en inglés y la presentación también, eh, Aitor y yo... Ο Άρτουρ και εγώ θα κάνουμε την παρουσίαση στα ε, ισπανικά, παρότι οι διαφανίες μας είναι στα αγγλικά. Σε 10 λεπτά λοιπόν θα παρουσιάσουμε κάποιες από τις ιδέες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ε, έκθεση. Δηλαδή θα αναφερθούμε, ε, στη, εγώ θα αναφερθώ πρώτα στο περιεχόμενο της ανάπτυξης ανθρωπιστικής βοήθειας ε, και τις ε, επιπτώσεις του Brexit και μετά ο Σέλφος θα μιλήσει για συγκεκριμένες περιπτώσεις και συγκεκριμένες επιπτώσεις της διαδικασίας. Εμείς θέλουμε ε, να αναφερθούμε στις ε, ενδεχόμενες επιπτώσεις του Brexit στις πολιτικές ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Θελήσαμε να δούμε το θέμα αυτό γνωρίζοντας ότι η έκθεση αυτή βρίσκεται ακόμα σε μεγάλη αβεβαιότητα, δηλαδή το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αβέβαιο. Ε, δηλαδή ε, εμείς προσπαθούμε να βρούμε κάποια εναλλακτικά σενάρια περιπτώσεων τις οποίες ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουμε ε, όταν προκύψει το Brexit. ένα έως 3% θα είναι, ε, είναι η συμμετοχή ε, της ε, Βρετανίας στην αναπτυξιακή βοήθεια και επομένως γι' αυτό ακριβώς κάπου εκεί θα βρίσκεται και ο αντίκτυπος. Ίσως μπορεί να υπάρξει και μια μείωση 10 με 30%. Εν πάση περιπτώσει όλα τα αριθμητικά στοιχεία θα πρέπει κανείς να τα ξαναδεί λαμβάνοντας υπόψη και την ε, αναγγελία μείωσης ε, της αναπτυξιακής βοήθειας από την πλευρά των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και εάν μάλλον λάβουμε υπόψη και τις γειτονικές χώρες προς την Ανατολική Ευρώπη και την Νότια Αφρική, ίσως τότε ο αντίκτυπος να είναι πολύ μεγαλύτερος με περικοπή της τάξης του 1 και έως και 4% ανάλογα με τα διάφορα σενάρια σενάρια. Ε, αυτά θα τα δούμε στις διαφορετικές προσεγγίσεις. Ε, εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι έστω και αν ε, η αναπτυξιακή πολιτική και η πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας δεν είναι ε, και από τα κεντρικά ζητήματα όσον αφορά την απόσυρση, ε, την αποχώρηση της, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της κατάστασης, ναι, μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι ο δωρητής του 50% της συνολικής βοήθειας. Είναι επομένως ε, ο πιο σημαντικός ε, δωρητής. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου που είχε κάνει και μια συμφωνία για το 0,7% του ποσοστού ΑΕΠ όσον αφορά την ανταξιακή βοήθεια που είναι σημαντικό ποσοστό λαμβάνοντας υπόψη την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου καταλαβαίνουμε ότι ε, είναι χώρα η οποία μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ε, ρόλο στα πλαίσια αυτού του γενικού ρόλου της Ενωμένης ΕΕ Ευρώπης όσον αφορά την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια και επομένως κατά αυτή την έννοια το Brexit θα μπορούσε να έχει σημαντική σημαντική διάσταση ας πούμε και θα πρέπει να συνυπολογιστεί στη συνολική, στο συνολικό Brexit ε, για να μπορέσουμε ε, ε, μάλλον εξ αρχής να πω ότι δεν έχουμε βεβαιότητες εδώ και επομένως εμείς κάναμε κάποιες παραδοχές έτσι ώστε να κινηθούμε σε διαφορετικά σενάρια. Πιστεύουμε ότι αυτή η μεθοδολογία είναι σημαντική έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια ε, συμπεράσματα. Ε, να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα λοιπόν τα οποία ε, να περιλαμβάνουν και συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμητικά στοιχεία κτλ. Ε, αυτές ε, οι υποθέσεις ε, περιγράφονται στο πρώτο τμήμα αυτής της διαφάνειας. Πρώτον δηλαδή ότι το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει, αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε να θεωρήσουμε δεδομένη την αποχώρηση. Και μετά έχουμε και άλλα σενάρια τα οποία αφορούν ε, την ε, οικονομική αποδέσμευση ε, και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή, Υποθέτουμε ότι το ΑΕΠ και των δύο πλευρών θα διατηρηθεί περίπου στο ίδιο επίπεδο μέχρι το 2020 περίπου. Αυτό είναι το ε, σενάριο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις του Brexit ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Βοήθεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΣΑ ακολουθούν περίπου την ίδια γραμμή σκέψης αλλά υποθέτουμε επίσης ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές ε, αλλαγές στην στα, ε, στα νομίσματα ε, λέμε ότι μπορεί να, υπάρξουν κάποια, να υπάρξει κάποια ε, υποτίμηση η, οποία δεν θα ξεπεράσει το 30%. θεωρούμε ότι στην περίπτωση ε, του Ηνωμένου ε, Βασιλείου ε, σύμφωνα με τις αναλύσεις που έχουμε κάνει δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιες παραμέτρους ιδιαίτερα πτυτικές ας πούμε και εναλλασσόμενες. Επίσης θεωρήσαμε σαν υπόθεση ότι οι δεσμεύσεις οι οικονομικές μέχρι το 2020 θα διατηρηθούν γιατί τότε λίγη συμφωνία του Κοτονού και γιατί τότε είναι το πιο πιθανό ότι θα γίνει η πραγματική έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, και επίσης γιατί το 20 ολοκληρώνεται ε, το πολιετές ε, πλαίσιο. Βασιστήκαμε λοιπόν πρώτα τον ε, προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεύτερον, ο τρόπος ε, με τον οποίο θα γινόταν η γεωγραφική κατανομή και πώς θα γινόταν η κατανομή ανά κάθε μέσο και επίσης τις δυνατότητες συνεργασίας μετά το Brexit μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως έλεγα και προηγουμένως, ε, αυτή η δέσμευση του 0,7% ε, είναι δεσμευτική νομικά. Ε, υπάρχουν βεβαίως κάποιες φωνές κατά αυτής της νομικής συμφωνίας, κάποιοι αντιτίθενται και το λένε που θα μπορούσε ε, ε, εάν ε, η δική τους πλευρά κερδίσει ας πούμε να μειωθεί κατά πολύ αυτό το ποσοστό. Αυτό θα γίνει λόγω εσωτερικών λόγων ή λόγω του ότι τελικά θα υπάρξει μια σημαντική υποτίμηση της λίρας στερλίνας. Πάντως ε, παραμένει η πιθανότητα να παραμείνει ακριβώς αυτό το συμφωνημένο ποσό στο 0,7 ε, και ε, μάλιστα χθε ε, η Υπουργό Ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου υπογράμμισε την ανάγκη να παραμείνει αυτό το ποσοστό τη ανθρωπιστική, τη αναπτυξιακή βοήθεια. Εμείς διατηρήσαμε το στοιχείο αυτό γιατί έπρεπε να βασιστούμε και σε ένα ε, ε, ε, ποσοστό συγκεκριμένο αριθμητικό. ε, βασιστήκαμε στο, στην υποτίμηση του 3, κατά 30% της λίρας. Αυτό είναι ένα, ένας μέσος όρος που μπορεί να αποτελέσει ένα λογικό ποσοστό που μπορεί να ακολουθήσει, να έχει μάλλον σαν επακόλουθο τη μείωση ανθρωπιστικής αναπτυξιακής βοήθειας αντίστοιχη με αυτήν που είδαμε από χώρες οι οποίες αντιμετώπισαν κρίση. Ε, στην Ισπανία είχαμε μονάχα ε, μια πολύ μεγάλη μείωση του 75% όσον αφορά την αναπτυξιακή ε, βοήθεια και αυτό είναι το μεγαλύτερο δυνατό. Επίσης μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις στο στρατηγικό μοντέλο βασιστήκαμε σε αναλύσεις που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε αναλύσεις ε, ε, του Brexit σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια και θεωρήσαμε ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες. Η μία πιθανότητα ε, θα μπορούσε να είναι ότι η βοήθεια μπορεί να ακολουθήσει ένα, ένα μορφότυπο πιο συγκεκριμένο. Επομένως, η, η βοήθεια η οποία δίνει δίνονταν μέχρι τώρα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον να δίνεται ε, μέσω διμερών συμφωνιών ε, της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης η γεωγραφική κατανομή θα εξαρτιόταν από τα διμερή προγράμματα και συμφωνίες μάλλον και ενδεχομένως σαν τομεακή ας πούμε κατανομή θα αφορούσε τις οικονομικές ε, τις οικονομικές ε, υποδομές ε, και εδώ θα ξανααναφερθώ εις την Υπουργό Ανάπτυξης η οποία αναφέρθηκε και υπογράμμισε ιδιαίτερος την ανάγκη συνέχισης των δεσμεύσεων και εμπορικών συμφωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η βοήθεια επίσης θα μπορούσε ε, ενδεχομένως να διατηρήσει και τον μορφότυπο της ε, ευρωπαϊκής και τα χαρακτηριστικά της ενωσιακής ε, βοήθειας. Γιατί ευθυγραμμίζεται σε πολλές περιπτώσεις και σε μεγάλο βαθμό η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρχές βάσει των οποίων δηλαδή δίνεται η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές της, του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα, εάν ακολουθήσει λοιπόν η βρετανική βοήθεια ε, αυτό το πατρόν, αυτό το μορφότυπο ας πούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε ε, θα συνεχίσει να δίνεται μέσα από τις, ε, τους ίδιους διάβλους και με την ίδια μορφή που έχει αυτή τη στιγμή και η ε, ε, ε, ενωσιακή βοήθεια. Υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση, δηλαδή να ακολουθήσει η Βρετανική βοήθεια ένα σχήμα το οποίο εμείς ονομάζουμε κοσμοπολίτικο ή παγκοσμιοποιημένο. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, θα ακολουθηθεί το ίδιο τομεακό και ε, γεωγραφικό ε, ε, σχήμα ας πούμε το οποίο θα προωθεί την βοήθεια μέσα πλέον από τα από διάβλους που θα ορίζονται μέσα από τις διμερείς συμφωνίες. Ε, ε, τώρα, για να προχωρήσουμε θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία περίπτωση ε, να εξακολουθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα και μετά από τον Brexit να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορεί και να ακολουθήσει την άλλη περίπτωση να μην συνεργάζεται μετά το Brexit. Αυτή είναι η τελευταία μεταβλητή. Εμείς σαν θεώρηση εργασίας είπαμε ότι θα ακολουθήσουμε τρεις υποθέσεις εργασίας τρία διαφορετικά σενάρια, ε, στα οποία όμως θεωρούμε δεδομένο ότι η εξέλιξη και από γεωγραφική άποψη και όσον αφορά του ε, διάβλους ε, κατανομής αλλά και όσον αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας θα είναι παρόμοια με αυτά και θα εξελιχθούν ομαλά επομένως όλες αυτές οι παράμετροι και θα είναι παρόμοιε με τι παραμέτρου που είχαμε δει μέχρι τώρα. Εμείς καθορίσαμε τα τρία σενάρια ως σενάριο εθνικιστικό, ε, ρεαλιστικό και κοσμοπολίτικο. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε αυτή την μείωση του 30% που έχουμε σημειώσει ήδη από την αρχή ε, το σχεδιάγραμμα ε, θα είναι ρεαλιστικό, δηλαδή θα ακολουθηθεί θα ακολουθηθούν τα διμερεί προγράμματα, η βοήθεια ε, θα δίνεται μέσα από οικονομικές δομές και στο σενάριο αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο ρεαλιστικό σενάριο παραμένουν τα χαρακτηριστικά, είναι τα ίδια χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες συνεργασίας ε, είναι μικρές ή μηδαμινές, αλλά διατηρείται ο όγκος της βοήθειας. Ε, αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί ως σενάριο γιατί η Υπουργός Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου Ε, υπογράμισε ε, ε, ότι, το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν φεύγει από όλο τον κόσμο και από όλες τις υφιστάμενες δομές και επομένως έχει την πεποίθηση ότι πρέπει να συνεχίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να, είναι, να παραμείνει δεσμευμένο κατά κάποιο τρόπο στρατευμένο στην αναπτυξιακή βοήθεια. Και η βοήθεια λοιπόν θα γίνει μέσα από τις ε, διάβλους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είτε συμμετέχοντας σε μηχανισμούς ταυτόχρονης παρουσίας και συνεργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό μπορεί να συμβεί όπως έλεγα και προηγουμένως γιατί πολλά από τα χαρακτηριστικά της βοήθειας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τις αντίστοιχες δομές του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς ότι θα, κράτη, θα διατηρηθεί ακριβώς στο ίδιο επίπεδο και με τους ίδιους ε, τρόπους και τα ίδια κανάλια ας πούμε και διάβλους ε, η, η βοήθεια από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, υπάρχει και το, το τρίτο σενάριο, αυτό που εμείς ονομάζουμε κοσμοπολίτικο, όπου η βοήθεια θα ακολουθήσει άλλες διάβλους μέσα από διμερείς συμφωνίες αλλά και εκεί θα υπάρξουν δυνατότητες ε, συνεργασίας ε, μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου σε ένα σενάριο post-Brexit, αφού δηλαδή εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά είναι τα σενάρια, αυτές είναι οι υποθέσεις εργασίας, τις οποίες εμείς θελήσαμε να αναπτύξουμε, βασιζόμενοι ακριβώς σε αυτές τις παραμέτρους που ανέφερα, έτσι ώστε να δούμε ποια μπορεί να είναι τα επιχειρημα μπορεί να είναι οι επιχειρησιακές, ε, επιχειρηματικές, οικονομικές, ε, εμπορικές επιπτώσεις του Brexit. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον συνάδελφο. Πολύ σύντομα θα σας δώσω και εγώ κάποια στοιχεία τα οποία ε, ακριβώς το παρουσιάζουν τις επιπτώσεις γιατί ε, γιατί και αυτά τα αναφέρουμε στην μελέτη μας. Βέβαια πρέπει να έχετε διαβάσει ε, άλλα στοιχεία πριν φτάσουμε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, όπως σας ε, είπε και η συνάδελφος, εμείς, εμείς δουλέψαμε με βάση τρεις υποθέσεις εργασίας, τρία σενάρια, τα οποία μπορεί να είναι το ένα πιο ρεαλιστικό, το άλλο πιο εθνικιστικό, το άλλο πιο κοσμοπολίτικο και βασίζονται βεβαίως στις πολιτικές αποφάσεις κλειδιά, τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα ε, ληφθούν στα πλαίσια της απομάκρυνσης του Ηνωμένου Βασιλείου από, το, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν βλέπετε αυτόν τον ε, πίνακα, αλλά εδώ βλέπετε σε εκατομμύρια δολάρια ε, αυτές τις επιπτώσεις. Εμείς ε, στην ποσοστοποίησή μας ε, χρησιμοποίησαμε ε, τα στοιχεία στατιστικής του ΟΣΑ. Ε, αυτά τα στοιχεία λοιπόν τα οποία χρησιμοποιεί όσα έτσι ώστε να λύσει προβλήματα τα οποία πολύ συχνά αποτελούν σημαντικό πρόσκομα στην ομαδοποίηση στοιχείων και δεδομένων. Ε, εμείς θελήσαμε να ακολουθήσουμε μια ενιαία ας πούμε γραμμή. Ε, είδαμε λοιπόν τα στοιχεία, τα βάση της ομαδοποίησης του ΩΣΑ έτσι ώστε να δούμε ε, ποια επίπτωση θα μπορούσε να έχει στην αναπτυξιακή πολιτική η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου. Και βλέπουμε ότι ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια δολάρια. Ε, στα 13, ε, από τα 13.670 στην κατάσταση πρώτου Brexit ενδεχομένως θα μπορούσαμε να φτάσουμε κάπου ανάμεσα από 11.30 και 12.30 ε, περίπου ανάλογα με το σενάριο το οποίο θα ακολουθηθεί. Βεβαίως εμείς ξεκινούμε με την ε, παραδοχή ότι ε, οπωσδήποτε θα υπάρξουν νέες ε, συμφωνίες, θα διατηρηθούν κάποια ποσά, αλλά ότι θα πρέπει να γίνουν συμφωνίες ανά περίπτωση και ανακλάδο. Όσον αφορά την συγκεκριμένη πολιτική. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη, είναι η εκρίζωση της ένδυας ε, και εάν ε, και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν εξακολουθήσουν να ε, προσπαθούν να καταπολεμούν αυτά, ε, αυτά τα προβλήματα, τότε οπωσδήποτε μπορούμε ε, να πούμε ότι ναι μεν θα συνεχιστεί η αναπτυξιακή αυτή η βοήθεια, αλλά οπωσδήποτε στο σύνολό τη θα είναι μικρότερη, γιατί, αλλά θα μπορούσε να έχει ένα αντίκτυπο της τάξης του 3% που σημαίνει ότι δεν είναι και κάτι τρομερό. Τώρα, ε, η ενδοξιακή βοήθεια δεν αναφέρεται μονάχα στους στόχους της ανεπτυξιακής ε, βοήθειας αλλά ε, και στην παρουσία μιας δύναμης, στη δυνατότητα επιρροής και επομένως υπάρχουν και άλλα στοιχεία και αριθμοί που μας ενδιαφέρουν. Ας πούμε πόσο ε, μειώνεται το βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη συνολική αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη αποτελούν, αντιπροσωπεύουν λίγο παραπάνω από το 50% της συνολικής βοήθειας και επομένως εάν φύγουν, αν φύγει η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου προφανώς δεν θα φτάσουμε σε αυτό το 50%. Ε, και οπωσδήποτε αυτός ο αριθμός του 50% και πάνω της συνολικής αναπτυξιακής βοήθειας που δίνεται από την ε, από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως αναφέρθηκε ε, στη δήλωση για την κατάσταση της Ένωσης, προφανώς ε, μετά από το Brexit δεν θα είναι δυνατόν να καλυφθεί. Επίσης, να μην λησμονούμε ότι στην κατάσταση πριν από το Brexit το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πολυμερές σύστημα φτάνει στο 61% και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν θα επιτευχθεί. Ε, επίσης, όσον αφορά τις γεωγραφικές ε, περιοχές, ε, είναι πιθανόν να υπάρξουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την γεωγραφική κατεύθυνση των κονδυλίων. Ε, υπάρχουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα, οι χώρες της γειτνίασης, του συστήματος ε, ε γειτονίας που ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση του Brexit θα τροποποιηθούν. Στο πέμπτο τμήμα της ε, μελέτης ε, αναφέρουμε πολιτικές, οικονομικές, επιχειρησιακές επιπτώσεις ε, και εδώ θα δείτε και μια σειρά από διαφάνειες βάσει των οποίων προσπαθούμε να δούμε ποιες, είναι ή ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτές τις επιπτώσεις και απέναντι στη διπλή επίπτωση δηλαδή έξοδο της Ευρωπαϊκής, ε, έξοδο ε, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι απλή. Οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να αφήσουν ε, το, ε, τα, τα ποσά ε, ακριβώς εκεί που θα έχουν μείνει όταν θα έχουν αφαιρεθεί τα ποσά του Ηνωμένου Βασιλείου ή ε, έχουν την δυνατότητα να προσπαθήσουν να αυξήσουν ε, την βοήθεια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να αντισταθμιστεί η εχουν την δυνατοτητα να προσπαθησουν να αυξησουν την βοηθεια απο Βεβαίως, η συνολική στρατηγική ε, της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης θέλει να διατηρήσει αν όχι να αυξήσει τον ίδιο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως βεβαίως θα εξακολουθήσει να θέλει να υπογραμμίσει κυρίως τις προτεραιότητες όσον αφορά της, την γειτονία, της χώρες γειτονίας. Βεβαίως ε, θα πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πόσον ε, στην ε, νέα διαμορφωθήσα κατάσταση, εάν θα θέλει μόνο να παραμείνει στις παλαιές προτεραιότητες γειτονίας ή αν θα θέλει να, να διασφαλίσει τον ρόλο του συνολικού ας πούμε παίχτη. Ε, από την άλλη πλευρά, ε, ε, ακόμα και σε περιπτώσεις του εθνικιστικού σεναρίου ή και του ρεαλιστικού σεναρίου από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδεχομένως θα, χρειαστούν, θα χρειαστεί αύξηση των πόρων. Εν πάση περιπτώσει, σε κανένα από τα σενάρια αυτά δεν περιμένουμε αντιστάθμιση της απώλειας του 15 100 της ε, χρηματοδότησης. Ε. Ε, μάλλον μπορούμε να αναμένουμε μια επανοργάνωση από γεωγραφική άποψη. Όσον αφορά τώρα τις πολιτικές επιπτώσεις, νομίζω ότι η ανάγνωση θα είναι περίπου ίδια στο εθνικιστικό σενάριο ας πούμε, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, αποφασίσει αύξηση του συνολικού ποσού, ε, πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει επανεστίαση της γεωγραφικής ε, κατανομής. Ε, εάν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θελήσει να, έχει, να ακολουθήσει ένα προφίλ περισσότερο περιφερειακό και όχι τόσο συνολικό τότε αυτό το 15% της απώλειας των πόρων ε, θα ε, ήταν επιζήμιο στην ουσία ε, για τις χώρες της Αφρικής ή της Καραϊβικής γιατί θα εξακολουθήσει να είναι, να είναι προτεραιότητα ή να είναι προτεραιότητα οι χώρες της γειτονίας. Τέλος, έχουμε ένα τελευταίο τμήμα όπου αναφερόμαστε στη μελέτη μας, όπου αναφερόμαστε ε, στις ε, επιχειρησιακές ας πούμε διαστάσεις ε, ή εκφάνσεις της πολιτικής, τον τρόπο με, τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται τα κονδύλια, ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεται με τους διάφορους φορείς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτό, δηλαδή ε, μπορούν να υπάρχουν διαφορετικά σενάρια ή μάλλον διαφορετική διάβλη επικοινωνίας μέσω διμερών σχέσεων, μέσω πολυμερών σχέσεων ή μέσω συνεργασίας με μη κυβερνητικού ε, φορείς. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι σε γενικές γραμμές το ίδιο ποσοστό ε, και το, η ίδια ανάμειξη εργαλείων που χρησιμοποιεί τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να προωθήσει την ε, βοήθειά της θα εξακολουθήσει να υπάρχει, να υφίσταται και μετά από τον Brexit. Βεβαίως ενδεχομένως θα υπάρξει, μάλλον προτίθεται το ερώτημα κατά πόσο θα υπάρξει μία μείωση σχέσεων με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις της Βρετανίας και αν θα υπάρξει και μία μείωση της επιχειρησιακής ε, ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εμείς λέμε ότι και στις δύο περιπτώσεις ε, δεν θα προκύψει ιδιαίτερη μείωση της ικανότητας. Ολοκληρώνεται η εργασία μας με μία σειρά συστάσεων ε, οι οποίες αναφέρονται ακριβώς σε αυτή την συγκυρία που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να παραμείνει ε, global actor ε, και να εξακολουθήσει, αν θέλει δηλαδή να εξακολουθήσει να έχει αυτόν τον παγκόσμιο ρόλο και εκεί θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της ή αν θέλει να παίξει περισσότερο περιφερειακό ρόλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αναφερθήκατε και σε συμπεράσματα και σε στάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς διαπραγματεύσεις θα γίνουν, τι επιλογές θα θέσει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τι θα πούν ε, οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά για πολλές από τις υποθέσεις που κάνετε. Να δώσω λοιπόν το λόγο καταρχάς στον Σαρλ Γκέρενς που είπα για όσους ε, δεν ήταν εδώ, ότι θα είναι το σημείο επαφής μας, ε, τη επιτροπή μας για το Brexit, από εδώ και στο εξή. Σαρλ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω παραθέτοντα τον Γιώσεφ Λούντς, που είναι πρώην Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν ε, του, της Ολλανδίας ε, την επόμενη μιας ε, σχηματισμού ενός κυβέρνησης όταν είχε ενισχυθεί πάρα πολύ ο Υπουργός Εξωτερικών είχε πει το εξής όσο περισσότερο μειώνεται η επικράτεια ενός κράτους, τόσο μεγαλύτερος είναι ο εξωτερικός κόσμος. Το ίδιο συμβαίνει και με ε, την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο υπόλοιπο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος. Ε, δεν θα αλλάξουν πολλά, λένε κάποιοι, με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάνουν λάθος τα πάντα θα αλλάξουν και οι πολιτικές συνέπειες θα είναι σημαντικές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που ήταν η πιο πιστή όσον αφορά τη μεταγραφή στην πράξη των ε, δεσμεύσεων που είχε αναλάβει και ως προς τη χρηματοδότηση και ως προς την αναπτυξιακή πολιτική ε, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 7% ε, και αυτή η απώλεια θα είναι μεγάλη, δηλαδή θα μειωθεί η δυνατότητα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι μια τεράστια πολιτική συνέπεια όσον αφορά την ε, ισορροπία, τον συσχετισμό των δυνάμεων, για να το πω έτσι. Ε, είναι μια εξέλιξη η οποία είναι αντίθετη με το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, βάσει της οποίας έπρεπε να υπάρχει σύγκληση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Εδώ λοιπόν είδαμε, μας εξήγησαν όλες ε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ε, ε, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι φωτός απέχουμε από τις δεσμεύσεις που είχαμε θέσει πριν από πολλά χρόνια. Δεν καταφέρνουμε να είναι πλέον υποχρεωτική, ε, να είναι υποχρεωτικό ο χάρτη πορεία με την, το, την γραμμική πορεία που είχαμε προδιαγράψει μεταξύ του 2015-2030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 Φτάσαμε στο 0,7%. Ε, θέλουμε να φτάσουμε στο 0,7% μέχρι το 2030. Λέμε ότι 0,02% πρέπει να αυξάνεται ε, κατέτος η βοήθεια. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει καμία χώρα που να έχει επιτύχει αυτό το στόχο ε, που να κάνει αυτή την προσπάθεια με τον τρόπο με τον οποίο μόλις εξήγησα. Οπότε έχουμε χάσει δύο χρόνια ήδη από τότε που έγινε η διακήρυξη της της ε, Αιθιοπίας. Πέρα λοιπόν από ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πρέπει ε, να δούμε και τις υπόλοιπες συνέπειες του Brexit ε, στην αναπτυξιακή βοήθεια. Όταν θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο θα χάσουμε έναν καθαρό εισφορέα. Παρά ε, το, την επιστροφή των χρημάτων που τους επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 6 δις ε, ευρώ επιστρέφει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσουμε μία καθαρή εισφορά ε, περίπου του ίδιου επίπεδου. Τα κράτη-μέλη που διαπραγματεύονται τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δείτε τι θα γίνει του επόμενους προϋπολογισμούς. Η πολιτική ανα αναπτυξιακής βοήθειας ε, θα έρθει σε ανταγωνισμό με την κοινή γεωργική πολιτική, με τις ε, επιχορηγήσεις που περνάνε από τα διαρθρωτικά ταμεία. Οπότε θα προσπαθήσουμε ε, για όσους δεν συμφωνούν μαζί μας και για όσους η ανάπτυξη έχει απλώς μία ε, μειωμένη ε, σημασία. Για όλους αυτούς λοιπόν η πολιτική αναπτυξιακη βοηθεια θα είναι μία μεταβλητή προσαρμογή των άλλων πολιτικών. Δεν θα μου πείτε βέβαια ότι τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να αυξήσουν τα έξοδα, τις δαπάνε τους ως προς τον τομέα αυτό, ενώ όλοι όσοι βλέπουν ε, ε, την, τα, τα, τα έσοδά τους να αυξάνονται, ε, μπαίνουν στην κατηγορία των χωρών που ε, λανθασμένα που καλούμε καθαρούς ε, εισφορείς, γιατί περισσότερα παίρνουν και λιγότερα δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμένα λοιπόν με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Τα σενάρια hard Brexit, ε, σκληρό Brexit ή ήπιο, Brexit, δυστυχώς δεν μπορώ να διαβάσω το... δεν μπορώ να κάνω χειρομαντία για να ξέρω, δεν διαβάζω τον καφέ, δεν τα ξέρω όλα, όμως πρέπει να έχουμε μια κοινή θεώρηση ε, του τι ε, θα συμβεί ε, με την αντιπροσωπεία της Βουλής των Κοινοτήτων. Θα είναι λοιπόν αποδυναμωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε λιγότερα μέσα και τι θα γίνει με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω εμβασμάτων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη. Θα καταφέρουμε σε μια βραχυπρόθεσμη περίοδο σε μεταβατικό επίπεδο να πείσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεισφέρει μέχρι το τέλο του προγράμματο ε, με τι εθνικέ ε, ε, εισφορέ. Δεν νομίζω, δεν μου φαίνεται και πολύ σίγουρο αυτό, στο πλαίσιο των καταπιστευμάτων, των εισφορών των κρατών μελών που προστίθενται στις εισφορές της Επιτροπής θα μας λείψουν τελικά οι ε, εισφορές του Ηνωμένου Βασιλείου με κίνδυνο ε, επαναπροσαρμογής ε, των προγραμμάτων στις χώρες υπονάπτυξης. Λοιπόν, χαόδης θα είναι η κατάσταση, ένα μπάχαλο και συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτό τον όρο, αν ήταν χώρε οι οποίε ήταν ε, μικρή σημασία από απόψη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είχαν αποφασίσει να αποχωρήσουν, θα ήταν πολύ λιγότερο δραματική κατάσταση. Υπάρχει και ένα νεολογικό ζήτημα. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποια θα είναι η μελλοντική ε, ε ιδέα που θα έχουμε για την αναπτυξιακή πολιτική, αν ισχύσει το σενάριο που θα παραμείνει εταίρο σημαντικό στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα στον τομέα της πολιτικής ε, για τις χώρες ΑΚΕ. Σε αυτή την περίπτωση το Ηνωμένο Βασίλειο ε, που τότε θα είναι ένα εξωτερικό μέλος βέβαια, η άποψή του θα είναι πολύ σημαντική ίσω και περισσότερο από την χώρα, από μια χώρα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να βρούμε ένα κοινό έδαφος στο οποίο μπορούν να, το οποίο μπορούν να αποδεχθούν οι Βρετανοί. Ε, μέχρι τώρα υπήρχε μια καλή, ε, μια πολύ λογική προσέγγιση σε όλα και ήταν και πολύ πραγματιστική αυτή η χώρα. Δεν υπήρχε καμία πιο πραγματιστική χώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτή τη χώρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πολιτική, την αναπτυξιακή. Πώ θα το κάνουμε όμω αυτό, πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική αποδυνάμωση ε, και τη μείωση τη αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, πραγματικά Κάθε φορά το επαναλαμβάνω αυτό, αν όλες οι χώρες ε, έπρεπε να, ε, αν είχαν ε, επιτύχει τους στόχους τους του 0,7% σε 3-4 χρόνια, θα ήμασταν στο ίδιο επίπεδο εκταμιεύσεων που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή με το, Ευρωπα... με το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε τέσσερα χρόνια υπήρχαν και νέε εκταμιεύσεις και θα μπορούσαμε να το κάνουμε και χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι λοιπόν υπόθεση πολιτική, είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Ε, ε, θα πρέπει να ανασκουμποθούμε λιγάκι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να το διατυμπανίσουμε αυτό το πράγμα και θα πρέπει να επισημάνουμε τις αρνητικές συνέπειες και να έχουμε μια πολιτική αντίδραση πάρα πολύ σωστή και πολύ προσαρμοσμένη. Ε, νομίζω λοιπόν ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να κάνουμε και όσοι λένε για την εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω αυτή τη πολιτική αναπτυξιακή μεταφράζεται σε πράξη ο ευρωπαϊκό ανθρωπισμό. Δεν είναι λοιπόν εύκολο θέμα αυτό και είναι πραγματικά μεγάλη προτεραιότητας για όλους μας, ε, πρέπει πέρα από την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Ανάπτυξης, να αποστείλουμε ένα πολύ χειρό μήνυμα, να μην περιμένουμε πάρα πολύ, γιατί δύο χρόνια διαπραγματεύσεων περνάνε πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να είμαστε σαφείς ως θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα προ ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, πρέπει να το πούμε από τώρα. Ευχαριστώ πολύ για την επισκόπηση των διάφορων ζητημάτων και τη σοβαρότητά του και συμφωνώ μαζί σα μόλι βγήκαμε από μια συνεδρίαση που μιλούσαμε για μια νέα συνένεση. Υπάρχει ένα αισιόδοξο σενάριο σύμφωνα με το οποίο τα κράτη-μέλη θα αναπληρώσουν το κενό αυτό στη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι διαφαίνεται στη μελέτη σα. Αλλά αυτό δεν είναι το μήνυμα που, ακου... που ακούσαμε. Ε, Ξέχασα να πω το εξή. Είχε πει ο κύριο Πέρε ότι μία από τι επιλογέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ε, δώσουμε προτεραιότητα σε κάποιε περιφέρειε. Ε, ε, τι γίνεται όμω λοιπόν με το δόγμα των εξωτερικών σχέσεων τη κυρία Μογκερίνη, η οποία ενίσχυσε την πολιτική βούληση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα διεθνή ε, παίκτη. Βλέπετε λοιπόν ε, τι εικόνα θα δημιουργηθεί και οι ανησυχίε, οι φόβοι που θα δημιουργηθούν από όλε αυτέ τι συζητήσει. Εντάξει, Μέχρι στιγμής έχουμε δύο βουλευτές, τον Ενρίκε Γκενέρο, άλλοι μπορούν να προσταθούν, μπορούν να ζητήσουν να εγγραφούν στην γραμματεία. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Στο τέλος είχα μία ιδέα η οποία επηρεάζει πολύ συγκεκριμένα τι διαπραγματεύσει μα για τη συνένεση. Δημαχόμαστε για αυτό το 0,7% αλλά το επιχείρημα τη μεγάλη Βρετανία δεν το συζητήσαμε. Ίσως θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε τη δική μας επιχειρηματολογία. Τώρα ως προς την παρουσίαση θα έλεγα πως δεν μπορούμε παρά να μαντέψουμε τι θα σημάνει το Brexit για την αναπτυξιακή συνεργασία. Θα χάσουν τρεις παίκτες. Ο ένας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζητήματα αναπτυξιακής συνεργασίας θα χάσει πολιτική σημασία και αποδοτικότητα. Ο δεύτερος χαμένος είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή στο μέλλον είναι πολύ πιθανόν να είναι πολύ απομονωμένο στην αναπτυξιακή βοήθεια και το τρίτο, ο τρίτος χαμένος είναι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίοι θα έχουν λιγότερες δυνατότητες υποστήριξης ή και βοήθειας. Επειδή φυσικά όλα είναι πολύ ασαφή ακόμα. Δεν λάβατε υπόψη έναν τομέα αλλά πιστεύω πως πρόκειται για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία έχουν άμεσες επιπτώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να συμμετάχει, να έχει οικονομικά αν ακόμα και αν το 2019 γίνει το Brexit επειδή το δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να πληρωθεί από την Ευρωπαϊκή από το Ηνωμένο Βασίλειο στο 2020. Και επίσης πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για προγράμματα τα οποία συνεχίζουν μετά το 2020. Και πιστεύω πως αυτό πρέπει να υποθεί και να υπενθυμίζεται κάθε φορά εκ νέου στους διαπραγματευτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Επειδή έχουν υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορούν να διακόψουν μετά το 2019. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα είναι πώς θα είναι οι σχέσεις μετά θα υπάρξει μια δυνατότητα συνεργασίας ή, το Ηνωμένο Ασύλιο θα κινηθεί προς μια κατεύθυνση στην οποία θα προσπαθεί αυτή η καλή συνεργασία που είχαμε με την Κοτινού θα δημορφωθεί κατά τρόπον ώστε να απευθύνεται περισσότερο στην κοινοπολιτεία. Πιστεύω πως είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε οπωσδήποτε. Για εμάς και για τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές πιστεύω πως είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί αυτό που είπε και ο Σάρλς. Στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε το ΕΒ όσο το δυνατόν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούμε να σώσουμε οτιδήποτε σώζεται στη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Γκερέρο. Ε, ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο και θα κάνω ένα αστείο για την ε, Βρετανική παρουσία ε, στο ε, Προεδρείο με, το, με την Αν και τη Λίντα, αλλά τελικά δεν θα το κάνω το αστιάκι, γιατί είδα ότι εμείς οι Ισπανοί είμαστε περισσότεροι. Έχουμε και στη γραμματεία, έχουμε και στο πάνελ, έχουμε και κάτω. Επομένως, ε, επομένως εδώ μάλλον θα πρέπει να μιλήσουμε για την ισπανοβρετανική επιρροή επί του θέματος. Εν πάση περιπτώσει, ε, ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εργασία, έκθεση δυνατή και περιεκτική ε, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει ε, απέναντι στην διαπραγμάτευση ε, για το θέμα να, μελετήσουμε και το θέμα αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τι επίπτωση έχει το Brexit σε κάθε μία από τις εκφάνσεις και τους τομείς που μας απασχολούν και επομένως σε τέτοιες εργασίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όπως είπε λοιπόν ε, και ο Λιβιέ προηγουμένως ε, βεβαίως εδώ μιλάμε για σενάρια, ε, μιλάμε για πολλαπλές μεταβλητές τις οποίες ακόμα αγνοούμε και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτές τις μεταβλητές. Αυτό είναι το ένα μου σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο. Προσυπογράφω αυτά που είπε ο κύριος Γκέρενσε, κυρίως όσον αφορά την έμεση ή μία ας πούμε χρηματοδοτική οικονομική επίπτωση που θα έχει ε, στην αναπτυξιακή πολιτική και ε, ε, η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου. κοιτάξτε, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πάντα ε, δεσμευμένο, στρατευμένο στην ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Ακούγεται ότι ε, και επίσης ακούγεται ότι η Υπουργό Ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν πάντα ένα από τα σημαντικά στοιχεία των αναπτυξιακών συμβουλίων και αυτό το κεφάλαιο θα χαθεί. Ε, και βεβαίως ε, ο, ε, η επίπτωση μιας τέτοια απώλεια, ας πούμε, μιας τέτοιας υποχώρησης δεν μπορεί να μετρηθεί, είναι δύσκολο να μετρηθεί αλλά οπωσδήποτε θα είναι αρνητική σε σχέση με την ρόμη της αναπτυξιακής πολιτικής και αναπτυξιακής ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι στην πρώτη φάση τουλάχιστον, μάλλον το εθνικιστικό σενάριο ε, θα πάρει το πάνω χέρι. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον, το επίθετο εθνικιστικό γιατί τα πρόσημα είναι διαφορετικά και μας οδηγεί σε άλλες σκέψεις. Αλλά ας πούμε ότι θα είναι ένα σενάριο εντός του οποίου το Ηνωμένο Βασίλειο ενεργεί για τον εαυτό του, για το δικό του συμφέρον. Δεν ξέρω ε, εάν η Ιλιάνα ή ο Αϊτόρ μπορούν να με βοηθήσουν σε αυτό, αλλά ε, το αφήγημα της ε, Τερέζα Μέη έχει δύο στοιχεία που είναι από τη μία ας πούμε τα σύνορα και η μετανάστευση και η άλλη είναι ότι ε, θέλουμε να ε, ε, είμαστε πλέον αυτόνομοι, ανεξάρτητοι όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Δηλαδή υπονοείται ότι πλέον εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάψει το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει δεμένα τα χέρια από τις εμπορικές οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως θα ξαναγίνει μεγάλη δύναμη και θα γίνει περίπου η παλιά αυτοκρατορία που ήταν και πριν κάτι τέτοιο. Είναι γεγονός ότι σε μία πρώτη φάση πιστεύω ότι ε, η αναπτυξιακή βοήθεια θα χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο προώθησης εξωτερικής πολιτικής ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, τουλάχιστον στο πρώτο τμήμα, ε, γιατί μου φαίνεται ότι θα είναι πιο εγωιστική η αντιμετώπιση του Ηνωμένου Βασιλείου. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα ακολουθήσει το διεθνιστικό, ας πούμε, το κοσμοπολιτικό σενάριο. Εν πάση περιπτώσει, Δεν αρκεί να πούμε ε, ότι ενδεχομένως θα έχουμε σκληρό Brexit ή ελαφρύ Brexit ή μεσαίο Brexit ή ενδεχομένως καθόλου Brexit. Ε, αλλά νομίζω ότι ε, θα υπάρξουν διαφορές ανάλογα με το θέμα. Νομίζω ότι για την περίπτωση ας πούμε ε, της ελευθερίας μετακίνησης το Brexit θα είναι πολύ σκληρό ενώ για την περίπτωση ας πούμε των φοιτητών και των σπουδών θα είναι λιγότερο. Ευελπιστούμε ότι στην περίπτωση της αναπτυξιακής βοήθειας δεν θα είναι τόσο σκληρό το Brexit αλλά εμείς σαν Κοινοβούλιο και σαν Επιτροπή Επιτροπή Ανάπτυξης ε, θα πρέπει, θα πρέπει να ενεργήσουμε έτσι ώστε η, το, τελικό ας πούμε ε, ε, αντικείμενο ή αυτό που θα μείνει μετά από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου να είναι κάτι θετικό και κάτι φιλικό. δηλαδή να μην ξεκινήσουμε με αρνητικές σκέψεις και προθέσεις σε αυτήν την συζήτηση και διαπραγμάτευση για τα αναπτυξιακά. Να προσπαθήσουμε να βρούμε όσο γίνεται περισσότερους κοινού τόπους και όσο γίνεται περισσότερους κοινού παρονομαστές. Εν τέλει όμως αυτό που θα συμβεί θα εξαρτηθεί και από τους 27 Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρξει Brexit ε, και επομένως θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και οι 27 και να δουλέψουμε. Ε, και οι 27 θα πρέπει ε, να διατηρήσουμε λοιπόν το επίπεδο δεσμεύσεων που είχε το Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο όντως θα έπρεπε να αποτελέσει παράδειγμα για τους υπόλοιπους 27 γιατί με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική. Βέβαια ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και ποιο Brexit θα πέσει στο κεφάλι μας. Αλλά είναι βέβαιο ότι η έξοδος θα έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Θα υπάρξει μία πρώτη φάση όπου το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσπαθήσει να βάλει την αναπτυξιακή της ε, πολιτική στην υπηρεσία, της, ε, ε, υπηρεσία των, εξωτερικών της, των εξωτερικών του σχέσεων και εγώ φαντάζομαι ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο να ξεκινάει εμπορικά κέντρα, εμπορικές σχέσεις με πολλές χώρες σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ίσως κάνω λάθος αλλά εν πάση περιπτώσει τι να σας πω. στα χέρια μας είναι και μάλιστα ε, από τη στιγμή που ε, είμαστε 27 χώρες με δύο χεράκια η καθεμία, κάντε το λογαριασμό, πολλά χέρια προκύπτουν. Εν πάση περιπτώσει έτσι ώστε να μπορέσουμε, θα πρέπει να κινηθούμε όλοι έτσι ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο ε, που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, ε, είχε και την αναπτυξιακή βοήθεια, το τμήμα του και τη συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου. Δύσκολο το βλέπω να αυξηθεί η βοήθεια έτσι ώστε να αντισταθμιστεί το η μείωση, αλλά γιατί έτσι και είναι πολλά τα θέματα, δεν είναι μονάχα οικονομικό ε, ζήτημα, ε, πολλά άλλα παίζονται με την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λίντα. Εδώ έχουμε Ισπανούς, ε, αλλά έχουμε και αυτούς τους ξένους που μιλάνε και Ισπανικά. Άρα η Ισπανική παρουσία μεγαλύτερη. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τον Όρμπερτ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Είναι γεγονός ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και έχει δίκιο και ο Ενρίκε σε αυτά που είπε και ο Τσάρλς. Να μην λησμονούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, φεύγει μεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε, ήταν χωρισμένη η κοινή γνώμη. Ήταν και αυτοί οι οποίοι ήθελαν να, να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει να ληφθεί ε, η υπόψη και φαντάζομαι ότι ε, ε, ακριβώς επειδή είναι πολλοί αυτοί που συμφωνούσαν με την αναπτυξιακή βοήθεια έτσι όπως εδίνεται μέχρι τώρα, θα συνεχίσουν και μετά τον Brexit. Αυτό ελπίζουμε τουλάχιστον. Συμφωνώ, συμφωνώ και με αυτά που ε, ε, περιλαμβάνει η έκθεση. Βεβαίως, μη λησμονώντας ότι βασιζόμαστε σε ε, παραμέτρους αβέβαιες ε, και όπως είπε και ο Νόρμπερτ ε, θα πρέπει να δούμε κυρίως το σημείο 7 το οποίο, αυτό το 0,7 συγγνώμη το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε εν τέλει ε, ποιο σενάριο εν τέλει θα ακολουθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, ποιο θα είναι το πιο ρεαλιστικό σενάριο και ελπίζουμε ότι αυτό θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιους άλλους συναδέρφους που να θέλουν να πάρουν τον λόγο. Κάποιες ερωτήσεις όμως έχω. Σχετικά με τους αριθμούς που έδωσες. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να πιάσει το 0,7% έως το 2030 και φυσικά οι αριθμοί θα προσαρμοστούν. Έχετε βρει τι θα σημάνει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου συλλογικά για το 0,7% έως το 2030. Αυτό δεν ήταν σαφές. Επίσης πόσο μεγάλος χορηγός βοήθειας θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αν υποθέσουμε πως τα κράτη-μέλη δεν θα αυξήσουν μαζικά την βοήθειά τους όπως είναι και πιθανόν, όπως βλέπουμε σήμερα, και δεδομένων των οικονομικ... της οικονομικής συγκυρίας. Πόσο μεγάλος χορηγός βοήθειας, βοήθειας θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αλήθεια ότι είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Αν δεν τηρούσαμε τις ίδιες αναλογίες όπως σήμερα δεν θα ήταν αλήθεια. Κατάλαβα σωστά πως άλλες χώρες θα κάλυπταν το κενό στην περίπτωση του εθνικιστικού σεναρίου για μετά τον Brexit και της μη συνεργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου τότε θα έχουμε μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι σε ποια βάση το είπατε. Ήταν αρκετά αισιόδοξη πιστεύω. Και κάποια σχόλια ακόμα. Ακούγοντας τους συναδέλφους. Εάν σκεφτείτε πως συζητούμε για τη νέα συνένεση για το 2030, το, η παλιά συνένεση του 2005 συμφωνήθηκε υπό την Προεδρία του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τότε είχαμε την εκστρατεία του να κάνουμε τη φτώχεια παρελθόν. Και τότε είχε καθοριστικό ρόλο το Ηνωμένο Βασίλειο στο να επιτευχθεί η συνένεση αυτή του 0,7%. Έτσι με την αποδοτικότητα που επιτεύχθηκε με την πολύ σημαντική βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου την τελευταία δεκαετία. Παρά τις διάφορες κυβερνήσεις που υπήρχαν εκεί. γι' αυτό και πιστεύω πως στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε τον μόνο Υπουργό Ανάπτυξης που δεν υπόκειται στο Υπουργείο Εξωτερικών ή σε κάποιο άλλο Υπουργείο, όπως συμβαίνει στα περισσότερα άλλα κράτη. Έχει δηλαδή μια ισχυρή θέση στο Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο σε αντίθεση με άλλες χώρες, οπότε μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή. Αν δούμε λοιπόν τις πρακτικές συνέπειες της πολιτικής, θα δούμε στο τέλος πως ναι, ναι, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Πολλοί συναδελφοί είπαν πω μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να πάρει την απόφαση να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα έχει νόημα για την πρόοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει νόημα να συνεργαστούμε επί τη βάση τη συνεργασία με αναπτυσσόμενε χώρε. Και έχει νόημα επειδή συμμεριζόμαστε πολλέ κοινέ αξίε. Αλλά το τι θα γίνει απομένει να το δούμε με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο, κάποια τελική άποψη μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων, οπότε θα, περάσω, θα δώσω το λόγο στους ομιλητές. Δεν ξέρω ποιος θέλει να αρχίσει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια και τις ε, προτάσεις. Ε, εγώ θα ξεκινήσω με μια διευκρίνηση όσον αφορά ε, τη μεθοδολογία ε, που ακολουθήσαμε. Το επιχείρημά μας δεν είναι ότι η επίπτωση του Brexit ε, θα είναι μικρή στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Είπαμε απλώς ότι θα είναι περιορισμένο, όχι μικρή επίπτωση, περιορισμένη κυρίως ε, ε, περιορισμένη όσον αφορά ε, τα κονδύλια όσον αφορά δηλαδή, τη χρηματοδοτική συνεισφορά, επίσης περιορισμένη όσον αφορά την επιχειρησιακή δυνατότητα και τρίτον περιορισμένη επίπτωση όσον αφορά την πολιτική διάσταση σε σχέση με την επίδραση που μπορεί να έχει στην ε, στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ως δωρητών ε, και μέσω της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Βεβαίως, όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, δηλαδή την οικονομική επίπτωση, είναι εύκολο κανείς να υπολογίσει την οικονομική επίπτωση. Όταν αναφερόμαστε σε περιορισμένη επιχειρησιακή επίπτωση, λέμε ότι αντίθετα με άλλες πολιτικές ε, ε, ευρωπαϊκές ε, για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια δεν υφίστανται μεγάλα διοικητικά προσκόμματα σε συνεργασία ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, μετά από το Brexit. Γιατί αυτά τα καταπιστεύματα, τα trust funds, είναι, δίνουν την δυνατότητα τέτοια συνεργασία. Όσον αφορά την συμμετοχή ε, την συμμετοχή ε, ε, βρετανικών φορέων στο ευρύτερο σύστημα της Ένωσης για την ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή βοήθεια, ας πούμε μη κυβερνητικές οργανώσεις βρετανικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η συνεργασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά το Brexit. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με ε, διαφόρους και στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και επομένως δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι καλός μαθητής στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από τον Brexit όσον αφορά την αδεξιακή βοήθεια ή αν αντίθετα ακριβώς γιατί έχει επενδύσει ε, πολύ στην ε, αναπτυξιακή βοήθεια, μήπως ε, έχει πλέον την δυνατότητα, την αποτελεσματικότητα, την σαφήνεια στόχων έτσι ώστε να προχωρήσει μόνο του το Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίως είναι σαφές ότι δεν ήταν πάντα ο δωρητής ο οποίος περισσότερο ε, ε, διευκόλυνε ας πούμε τις γενικότερες ε, κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήταν δηλαδή η χώρα η οποία ήταν πιο εύκολη ας πούμε στην συνεργασία. Ε, ενδεχομένως λοιπόν αυτό οδηγήσει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κατά αυτή την έννοια και εάν ας πούμε διοικητικά ε, υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν πολλά εμπόδια αλλά είναι πολιτικά περισσότερο τα εμπόδια, εδώ ε, θα έχουμε έναν καλό δείκτη ε, του βαθμού στράτευσης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ε, όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Βλέπουμε όμως ταυτόχρονα, ταυτόχρονα δηλαδή με την εξέλιξη αυτού του προϋπολογισμού και αυτών των κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή, στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα μπορούμε να κάνουμε επομένως την σύγκριση με την εξέλιξη των προϋπολογισμών ε, των προπολογισμών των κρατών. Εκεί θα δούμε ότι οι τέσσερις έχουν μειώσει τον αναπτυξιακό προπολογισμό, αλλά τρει, η Ιταλία, η Γερμανία και η Σουηδία, έχουν αυξήσει ε, τον αναπτυξιακό τους ε, προϋπολογισμό. Και επομένως, μετά τον Brexit, είναι δύο οι δυνατές απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην νέα στην νέα κατάσταση. Είτε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίσει να συμπεριφερθεί ως ε, μία ε, περιφερειακή δύναμη η οποία θα βασίζεται στην ε, γειτονία ή και υπό την ηγεσία κάποιων συγκεκριμένων χωρών μελών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγηθεί προς μια άλλη κατεύθυνση και θα αποτελέσει επομένως έναν συνολικό ηγέτη. Όσον αφορά τώρα ε, πόσες είναι οι πιθανότητες το Brexit να είναι μαλακό ή σκληρό ή, ή μη σκληρό. Τώρα στις ε, επαφές που είχαμε και στις συνεντεύξεις ε, που ε, μας δόθηκαν, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, θα εξαρτηθεί από την συνεργασία και το βαθμό συνεργασίας που θα επιλεγεί μετά από το Brexit σε μια πολιτική ε, ε, πραγματικότητα το Brexit δεν γεννήθηκε ε, σαν αντίδραση προς την αναπτυξιακή βοήθεια. Επομένως θεωρούμε ότι δεν θα έχει μεγάλη μεγάλο αντίκτυπο και μεγάλη επίπτωση το Brexit στην αναπτυξιακή βοήθεια. Υπάρχουν άλλοι τομείς στους οποίους οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες. Απ' την άλλη πλευρά είναι ε, γεγονός και λαμβάνοντας υπόψη και την διάρθρωση των ε, ευρωπαϊκών ε, εργαλείων και μέσων, ενδεχομένως να είναι πολύ πιο εύκολη η συνεργασία μετά από το Brexit μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν έχει μεγάλη σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική το Brexit αν θα είναι πιο σκληρό ή πιο μαλακό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ. Ναι, θα προσπαθήσω να πω και εγώ δύο λόγια. Αυτό για το soft hard Brexit. Μπορούμε να το σκεφτούμε με την έννοια του πώς μπορεί να επηρεάσει τις μετέπειτα σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί, ας πούμε, εμείς σκεφτήκαμε ότι πολύ συχνά μας έλεγαν ότι πρέπει να σκεφτούμε τις ε, δυνατότητες που ανοίγονται, λαμβάνοντας ως ε, παράδειγμα την Ορβηγία και την ε, Σουηδία, οι οποίες είναι χώρες την Ορβηγία και την Ελβετία, συγγνώμη, οι οποίες είναι χώρες έφτα. Ε, ε, εμείς, ε, είδαμε και αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή το να γίνει το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, εν μια χώρα τύπου έφταλα αλλά εμείς θελήσαμε να δούμε περισσότερο μια, ένα πολιτικό σενάριο βάσει του οποίου το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να κρατήσει μια δικιά του πολιτική. Από την άλλη πλευρά, το Brexit Το Brexit ε, λέμε συχνά ότι ε, ε, σημαίνει ότι θα υπάρξει μείωση των πόρων των αναπτυξιακών κονδυλίων. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να συμβεί κάτι τέτοιο. και από την άλλη πλευρά δεν ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους ε, εάν θα ε, αυξήσει τα κονδύλια της αναπτυξιακής βοήθειας ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι να δούμε εάν τα χρήματα θα είναι τα ίδια και κυρίως εάν, θα, η διαχείρισή τους ε, θα είναι ε, παρόμοια. Σε ένα εθνικιστικό σενάριο το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε, αλλά αλλά και σιγά σιγά εγκαταλείπει και την θέση του στις διεθνείς υποδομές. Εμείς θεωρούμε ότι δεν ε, δεν θα είναι εύκολο να πάρει μια τέτοια θέση ε, η ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Εμείς πιστεύουμε ότι θα υπάρξει απλώς μια ε, μείωση ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου και τις οικονομικές, τους οικονομικούς περιορισμούς που υπάρχουν. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το ρεαλιστικό σενάριο. Ε, η αναπτυξιακή ε, πολιτική σχετίζεται με την εμπορική ε, πολιτική και επομένως δεν έχει λόγο να αλλάξει. Και να τελειώσω με κάτι άλλο που ρωτήσατε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κράτη-μέλη και ε, κομισιόν, ε, με ή χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, εξακολουθούν να είναι ο μεγαλύτερος δωρητής. Αλλά δεν θα ξεπεράσουν το 50% ε, της ε, βοήθειας. Η ταξινόμηση θα μπορούσε να αλλάξει των δωρητών μονάχα ε, σε, στην περίπτωση του εθνικιστικού ε, σεναρίου. Η, Κομισιόν ε, θα θα παραμείνει σύμφωνα με τα σενάριά μας στην τέταρτη σειρά, εκεί που είναι δηλαδή και τώρα, μετά από τη Γερμανία. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολλέ υποθέσεις γίνονται με λίγη βεβαιότητα. Νομίζω ότι τρία-τέσσερα συμπεράσματα μπορούμε να αντλήσουμε. Πρώτον, υπάρχουν ε, δύο λόγοι που εξηγούν ε, την αύξηση τη αναπτυξιακή βοήθεια. Πρώτον, η δέσμευση ε, των κρατών μελών στην αρχή τη δεκαετία του 70, η οποία ανανεώνονταν συνεχώς. Και δεύτερον, ε, είναι βέβαια η ανάπτυξη της, ε, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου που θα μας υποχρεώσει να ξαναδούμε από την αρχή την ε, ανάπτυξη, την αναπτυξιακή βοήθεια. Δεύτερο σενάριο που σημαίνει επικέντρωση ενδεχομένως στην άμεση, στις άμεσες γειτονικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν μου φαίνεται πάρα πολύ πιθανό, γιατί οι χώρες που βρίσκονται ανατολικά ε, είναι από μόνες τους έχουν μια συγκεκριμένη αναπτυξιακή βοήθεια. Η Ισπανία έχει παραδοσιακά κάποιες σχέσεις με την Αφρική. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Μου φαίνεται λοιπόν πολύ λίγο ρεαλιστικό αυτό το σενάριο. Το μόνο που μπορεί να μειώσει τον αριθμό των χωρών είναι ε, η αρχή της διαφοροποίησης την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όσο ε, ε, ε, σέβονται τα κριτήρια της ύπαρξης ενός μέσου εισοδήματος αποδεκτού, τότε εξαφανίζονται από τη λίστα των δικαιούχων της αναπτυξής βοήθειας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, ε, τρίτο σενάριο. Δεν νομίζω ότι το, Ευρω... το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξακολουθήσει να ε, διαχειρίζεται μόνη της ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, το λέω αυτό σε σχέση με όσα άκουσα κατά την ε, προεκλογική εκστρατεία ε, ε, κατά τη διάρκεια του, πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit. πάντοτε θεωρεί το ένα γραφειοκρατικό τέρας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ α, αμφιβάλλω ότι θα κάτσει το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθεί τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ αμφιβάλλω, μου επιτρέπετε. Εγώ έκανα λοιπόν αυτές τις παρατηρήσεις εν ώψη μια συζήτηση η οποία θα μας απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ του προσκεκλημένους ομιλητές μας για τις παρουσιάσεις τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μελέτη σας και για αυτά που μας είπατε. Είναι κάτι για το οποίο θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε. Ευχαριστούμε. It's food for thought and we'll watch this space. Πράγματι, μας έδωσατε πάρα πολλά πράγματα να σκεφτούμε. Mm-hmm. Πολλά ισπανικά ακούσαμε σήμερα και θα ακούσουμε ε, έχουμε τώρα την επόμενη συζήτησή μας ε, για τις σχέσεις της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική, σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης. Θα συζητήσουμε εδώ δύο πράγματα. Πρώτον, θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, ε, τον Ενρίκη Γκερέρο Σαλόμ, τη γνωμοδότηση για μια νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική. Πριν ακούσουμε όμως από τον Ερίκο από τον Ερίκη Γκερέρο, θα ακούσουμε ένα από τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Λατινική Αμερική και αυτό είναι το πρόγραμμα ε, Eurosocial, που είναι ένα πρόγραμμα ε, που, έχει, που είναι από τα βασικά μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής στην, στην Λατινική Αμερική. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στην ε, αναπτυξιακή βοήθεια της στη Λατινική Αμερική με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το κάνει στην Αφρική. Εξαρτάται από το είδος της κάθε χώρας ε, και τις συνθήκες. Είναι εδώ λοιπόν ε, ο κύριος Σαντομέ Καλέγη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Eurosocial και μετά θα ακούσουμε και την άποψη του Ενρίκη Γερέρο Σαλόμ. Δεν έχουμε συζητήσει τόσο πολύ το θέμα της Λατινικής Αμερικής όσο εγώ είμαι πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Είναι σημαντικό λοιπόν που σήμερα επικεντρωνόμαστε αυτό το σύντομα γιατί δεν νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει επαρκώς. Ακούμε λοιπόν τον Χουάν Μανουέλ Σαντομέ Καλιέχα, ο οποίος είναι διευθυντής ε, του ε, προγράμματος είναι ο διευθυντής του Eurosocial. Μπορείτε να μα πείτε εσεί περισσότερα για το πρόγραμμά σας. Ε, χαίρομαι που σα γνωρίζω. Καλώ ήρθατε. Μπορείτε να εξηγήσετε στου συναδέλφους. Πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν το πρόγραμμά σα. Μήπω μπορείτε να μα πείτε περισσότερα πράγματα. Έχετε γύρω στα 10 λεπτά στη διάθεσή σα. Και μπορείτε να μα πείτε πώ ταιριάζει με τη νέα αυτή στρατηγική είναι τμήμα όλη αυτή τη ε, διαδικασία. Καλό απόγευμα. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πρόσκληση. Χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας ένα, ε, συγγνώμη, ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το 2005. Και το διευθύνω ε, σχεδόν από την αρχή. Ε, άκουσα προσεκτικά αυτά που αναφέρατε προηγουμένως στη συζήτηση για τις επιπτώσεις του Brexit στις πολιτικές για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια και σκεφτόμουν ότι ε, είναι πάρα πολύ καλή η συγκυρία που τώρα εγώ πρέπει να σας παρουσιάσω ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς παρουσιάζει τα συγκεκριμένα αυτά χαρακτηριστικά και που μπορεί να ε, να δείξει ότι πέρα από την ποσότητα και η ποιότητα μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή δεν είναι μόνο το πόσα χρήματα ή πόσα κονδύλια έχει κανείς αλλά ε, και ο τρόπος που ε, κάνει την, την αναπτυξιακή πολιτική για οι επιλογές είναι κάτι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ε, κύριο πρωτοχικό σκοπό έχει την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής στην Λατινική Αμερική ε, και η συνοχή νοείται ε, και βάσει των αντικειμενικών αριθμητικών στοιχείων, μείωση των κενών και των ανισορροπιών, αλλά πρέπει να νοείται και ως ενδυνάμωση της κοινωνίας. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί πάνω από από 10 χρόνια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Λατινική Αμερική ε, ενισχύοντας ε, δημόσιες πολιτικές ε, για την κοινωνική συνοχή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο αντικειμενικά από άποψη αριθμητικών στοιχείων, αλλά είναι τεράστιο όσον αφορά ε, τις επιπτώσεις ε, που έχει. Ε, υπάρχει ένα κονσόρσιο Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας που είναι οι τρεις κεντρικές χώρες, όμως έχουν συμμετάσχει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ λοιπόν είχα προετοιμάσει για αυτά τα 10 λεπτά ε, κάποιες διαφάνειες, ε, ε, παρουσίαση λοιπόν κάποιων στοιχείων για να σας δείξω πού βρίσκεται ακριβώς η Νότια Αμερική σήμερα. Οι περισσότερες χώρες της Νότιας Αμερικής είναι χώρες μεσαίου εισοδήματος ή χώρες οι οποίες βρίσκονται στην μεταβατική περίοδο προς το μέσο εισόδημα και βεβαίως υπάρχουν εκεί και οι μεγάλες ε, χώρες όπως η Βραζιλία, η Χιλή, η Κολομβία κλπ. Ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας κάποια στοιχεία που αφορούν τη Λατινική Αμερική ε, έτσι ώστε μετά ε, να μπορέσω να μοιραστώ μαζί σας το πρόγραμμα, το πραγματικό πρόγραμμα του Eurosocial που αφορά την ανάπτυξη και την βοήθεια ε, να σας πω ότι πριν ε, λίγο πρόσφατα πήγαμε στο Παρίσι στην έδρα του ΟΣΑ ε, και το Κέντρο για την Ανάπτυξη του ΟΣΑ μας έλεγαν ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι, οι στόχοι του, ε, για το 2030 ακριβώς βασίζονται ε, στην γνώση, στην πραγματογνωμοσύνη, στις δημόσιες πολιτικές οι οποίες θα βελτιώσουν την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική συμπερίληψη. Εδώ θέλω να σας δείξω, ε, ξέρετε τον ε, δείκτη Gini, Εδώ έχετε λοιπόν ε, μία διαβάθμιση των χωρών ε, στην περιοχή, ε, ποιες έχουν μεγαλύτερο επίπεδο ανισορροπίας και ποιες όχι. Στη μία πλευρά έχουμε την Ουρουγουάη, στην άλλη έχουμε χώρες του τριγώνου της Κεντρικής Αμερικής. Μάθαμε ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να πάει ε, και σε αυτή την περιοχή. Η Ονδούρα και η Γουατεμάλα ε, είναι οι χώρες με, το, με την μεγαλύτερη ε, ανισορροπία και μιλάμε ε, για μια περιοχή με παραπάνω από 170 εκατομμύρια ε, ε, φτωχούς. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια τα οποία ζουν σε βαθμό τροτότητας πάρα πολύ μεγάλο και Είναι 217 περίπου αυτά τα εκατομμύρια ε, των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την κατάσταση που σας είπα και επομένως ο βαθμός τροτότητας αυξάνει και αναφερόμαστε εδώ ε, στην, ε, σε όρους ακραίας ή σχετικής φτώχειας, αναφερόμαστε στην πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση στην εκπαίδευση κτλ. Τα τελευταία χρόνια η Λατινική Αμερική ε, είδε το τέλος ε, ε, κάποιων χρόνων ανάπτυξης που ε, ακολουθήθηκε από την επιλογή αύξησης των δημοσίων ε, δαπανών. Ε, υπήρχαν τα χρήματα, ας πούμε, υπήρχαν τα αναπτυξιακά ταμεία τα οποία επέτρεψαν την αύξηση των δαπανών και που είχαν σαν αποτέλεσμα μείωση κάποιων ανισοτήτων και επίσης είχαν σαν αποτέλεσμα τη σχετική βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Ε, και σε γενικές γραμμές λοιπόν θεωρήθηκαν θετικό ε, εργαλείο. Είχαμε όμως την κρίση του 2010-2010 που είχε επίπτωση και στην ε, περιοχή. Επλήγει λοιπόν και η περιοχή από την κρίση αυτή. Μειώθηκε το ΑΕΠ Βλέπετε εδώ ταξινόμηση των χωρών ε, της ε, Λατινικής Αμερικής ε, βάσει της έλλειψης ισότητας και ισορροπίας. Εδώ βλέπετε ε, με το έντονο, ροζ, ε, έντονο σχέλ συγγνώμη, τις χώρες οι οποίες είναι πιο ε, αναπτυγμένες, Χιλή, Αργεντινή κτλ. Λοιπόν, εδώ ε, λέμε ότι το Ευρωσοσιάλ είναι ένα ε, πρόγραμμα το οποίο βελτιώνει την ε, κοινωνική κατάσταση γιατί οι ελλείψεις είναι πάρα πολλές. Μεταξύ αυτών η κεντρική θέση κατέχει το πρόβλημα της ισότητας των φύλων. Είναι 55% περίπου οι γυναίκες οι οποίες έχουν είτε καθόλου χρήματα είτε χρήματα πολύ λιγότερα από τους άντρες. Ε, ας πούμε στην Ονδούρα, στο Ελσαρβαδόρ και την ε, Γουατεμάλα, οι χώρες οι οποίες έχουν την χειρότερη, χειρότερη κατάσταση, ε, βλέπουμε εκεί μια σειρά στοιχείων όπως είναι η ένδια, η βία και επομένως εδώ πρέπει να βρούμε προγράμματα τα οποία θα δώσουν δουλειά στους νέους που θα βελτιώσουν την κατάσταση της δικαιοσύνης στη Γουατεμάλα ας πούμε όπου η κατάσταση όσον αφορά τη δικαιοσύνη είναι ιδιαίτερα ε, ευαίσθητη. Αλλά ε, Γουατεμάλα, Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, ε, Ονδούρα πρόκειται για χώρες οι οποίες και αποτελούν έτσι μέλημα της ΔΕΦΚΟ, της αρμόδιας υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το πλαίσιο ε, δεν είναι ακριβώς όπως το πλαίσιο της Αφρικής, αλλά υπάρχουν 15 χώρες οι οποίες ε, έχουν μεγάλα προβλήματα. Και γι' αυτό ακριβώς δημιουργείται το πρόγραμμα ε, Eurosocial το 2004 στο Μεξικό ε, στην τρίτη διάσκεψη κορυφής ε, Αμερικα... Λατινικής Αμερικής, Καραϊβικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλους αυτούς τους στόχους που έχω αναφέρει και προηγουμένως μείωση των ανισοτήτων, κοινωνική συμπερίληψη να, να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις εμπιστοσύνης έτσι ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική συμπερίληψη και έτσι ώστε να προκύψει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Εδώ θα σας δείξω έναν δικαστή Ισπανό και που θέλω να τον ακούσετε να περιγράφει το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να τον ακούσουμε. Yeah. No. Yeah, John said let her do it. Yeah. Yeah. Yes, Caroline. Yeah. Bueno, él es un magistrado que... En base περιπτώσει,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 para atacar y solucionar ese problema. Para mí, este último elemento es precisamente la singularidad de lo social. Sorry for that, I was just explaining that for those who didn't speak Spanish, there no interpreting for these videos, so not a good, it's difficult in committee. Έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η διερμηνία από βίντεο, λέει η Πρόεδρος, γιατί ο ήχος δεν είναι καθόλου καλός. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, την μαρτυρία ε, αυτού του δικαστικού. Είναι ένας δικαστής ο οποίος ε, συνεργάστηκε πάρα πολύ στην φάση 2 από το 10 μέχρι το 15 ε, και προσπαθούσε ακριβώς να εξηγήσει τα πράγματα και ε, ε, εξήγησε πάρα πολύ καλά τους στόχους του προγράμματος, τον τρόπο συνεργασίας, ε, ε, αυτήν την συνεργασία μεταξύ ε, ισοτήμων ανθρώπων του δημοσίου τομέα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευρά των χωρών της Λατινικής Αμερικής που προσπαθούν να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές έτσι, ακριβώς, έτσι ώστε ακριβώς να βελτιώσουν την κατάσταση, να βελτιώσουν τον διάλογο ε, με τρόπο ώστε να προκύψουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε κοινωνική συνοχή, κοινωνικές αλλαγές και βελτίωση γενικότερα του κλίματος σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Είναι πολλές ε, οι πολιτικές ε, ε, συνοχής ε, που είναι ιδιαίτερα προσφυλής ε, στην Ευρώπη. Πολλά έχει η Ευρώπη που μπορεί να μοιραστεί με τον υπόλοιπο κόσμο και επομένως και με τη Λατινική Αμερική. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είχαμε και μια πολύ καλή συνεργασία νότου-νότου, δηλαδή μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Κάθισαν γύρω από το τραπέζι Αργεντίνοι οι οποίοι μοιράστηκαν στρατηγικές ανάπτυξης με το Σαλβαδόρ ε, και τα λοιπά. Ε, ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά θα, δεν έχετε άλλο χρόνο στη διάθεσή σας. Άλλωστε έχουμε εδώ το πρόγραμμα. Πρέπει να αφήσουμε και χρόνο έτσι ώστε να μιλήσει και ο κύριος Γκερέρο. Εν συνόψη, να σας πω ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει ακριβώς να δημιουργήσει γέφυρε ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να βελτιωθούν τα προβλήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν προβλήματα τα οποία χρήζουν ε, καινοτόμων, έτσι, δημιουργικών πολιτικών ε, για να αντιμετωπιστούν και επομένως ε, έχουμε ακόμα πέντε χρόνια, θα συνεχίσουμε την συνεργασία, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κοινωνική συνοχή σε όλες τις περιφέρειες. Ευχαριστώ. Ε, uh, έχουμε σκοπό και εμείς να επισκεφθούμε την Κεντρική Αμερική και να δούμε κάποια από τα προγράμματα του Eurosocial. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που μας, είπε, που μας είπατε για την αναψυχική συνεργασία στη Λατινική Αμερική και τώρα θα δώσω το λόγο στον Ενρίκε Γκερέρο να μας πει ορισμένα πράγματα για τη δική του ε, έκθεση σε σχέση με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω και τον Χουάν Μανουέλ όχι για την ε, ε, έκθεση, την εισήγηση που μας έκανε εδώ, κυρίως να τον ευχαριστήσω για την δουλειά που έχει κάνει στην Λατινική Αμερική μέσα από την μεταφορά, ας πούμε, ε, της ευρωπαϊκής εμπειρίας, αλλά και μέσα από την σκληρή δουλειά που κάνει. Ήθελα να πω ότι η γνωμοδότηση που θα συζητήσει η Επιτροπή μας αφορά μία έκθεση της ε, ΑΦΕΤ ε, που έχει στρατηγικό χαρακτήρα και που ε, λέει ότι ε, πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Ε, από τη στιγμή που οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ξεκινήσει αυτό την οδό του απομονωτισμού και έχουν αρχίσει ε, να ε, αποκλείουν χώρες μεταξύ άλλων και της Λατινικής Αμερικής ε, δυναμητίζουν, θέτουν εν κινδύνο την οικονομία το πολλών χωρών μεταξύ των οποίων και το Μεξικό και αυτή ακριβώς είναι η κατάλληλη στιγμή, η απαραίτητη στιγμή έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει την ε, το κενό το οποίο ε, αφήνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε που άλλοι μπορούν να το βλέπουν θετικό και άλλοι αρνητικό. Εξαρτάται. Εμείς ακριβώς θέλουμε να ε, εντάξουμε την προοπτική της αναπτυξιακής βοήθειας και διέπεται η αρχή αυτή από κάποιες βασικές αρχές. Πρώτον, ότι η Λατινική Αμερική, όπως άλλωστε υπόθηκε, ε, είναι μία ήπειρος με πολύ υψηλό βαθμό ανισορροπίας. Δεύτερον, οι χώρες αυτές οι οποίες ε, και παρότι θεωρούνται μέσω εισοδήματος έχουν ε, εντός τους προβλήματα περιφερειακά, μειονοτήτων, ε, ε, ηλικιακά, φιλε, διακρίσεις φύλου κλπ. τα οποία ενέχουν ακριβώς και οδηγούν σε μεγαλύτερη ανισορροπία. Και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να έχει μια ισχυρή αναπτυξιακή σχέση με τις χώρες αυτές, όχι μόνο λαμβάνοντας υπόψη το μέσο εισόδημα των χωρών αυτών, αλλά μέσω ανάλυσης ε, αντικειμενικής ε, ε, της πραγματικότητας των χωρών αυτών, έτσι ώστε να ξέρει ανα πάσα στιγμή ποια είναι η ισορροπία την οποία καλείται να βοηθήσει. Όπως προτάθηκε προηγουμένως πρέπει να υπάρχει διάλογος, πρέπει να υπάρχει διαπραγμάτευση, πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες έτσι ώστε μέσω κοινών στρατηγικών χωρών λοιπόν Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν ε, η γνωμοδότηση θέτει κάποια ερωτήματα κάποια ζητήματα. Πρώτον, μεγαλύτερη σημασία στην διακυβέρνηση ε, και εδώ μπαίνει και η καταπολέμηση της ατιμορρησίας, ε, της ε, διαφθοράς, να διασφαλιστεί ένα μερόληπτο δικαστικό σύστημα, να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις της διοίκησης και ενίσχυση της διοίκησης. Είδαμε ότι υπάρχουν χώρες μας, τις παρουσιάσατε προηγουμένως, ότι υπάρχουν προβλήματα διακυβέρνησης, ε, ε, χώρες ε, με μεγάλη βία, χώρες οι οποίες είναι σχεδόν fail states και επομένως αυτά θα πρέπει να τα μιλήσουμε, να τα αναφέρουμε. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε για ενίσχυση των δημοσίων πολιτικών που παρέχουν ευκαιρίες εμπορικές συνεργασίας κλπ. Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές κινήσεις εμπορικές, οι οποίες όμως από μόνες τους δεν μπορούν να φέρουν αυτήν την κοινωνική ισορροπία, την κοινωνική ε, συνοχή και επομένως θα πρέπει να ενισχυθούν δημόσιες πολιτικές στην υγεία, στις ε, υποδομές, στην κοινωνική πολιτική, στην εκπαίδευση κλπ. Επίσης, λέμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα ε, εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να επιδιωχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με βεβαίως ε, προαγωγή ε, και σεβασμό και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών κτλ. Θέλουμε να υπάρξει διάλογος μεταξύ των συνδικάτων, μετά τη συνδικαλιστικής οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Να προαχθεί λοιπόν ο διάλογος, να ε, ληφθεί λαμβανθεί υπόψη επίσης η κλιματική ευαισθησία των χωρών αυτών. Ε, όλη η περιοχή της Καραϊβικής αντιμετωπίζει ισχυρό κλιματικό ε, κίνδυνο κυρίως για το μέλλον αλλά ήδη τώρα γνωρίζουμε και στην Επιτροπή μας ότι όλο και περισσότερο ε, υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες κλιματικοί για λόγους δηλαδή αλλαγής κλίματος. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, ε, οπωσδήποτε να δοθεί σημασία στην ε, διακριτική μεταχείριση των γυναικών, διακρίσεις λοιπόν που οφείλονται στο φύλλο ε, και να θυμίσουμε επίσης ότι Υπάρχουν ε, στοιχεία όπως ε, η συνοχή των πολιτικών, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην εμπορική και την αναπτυξιακή πολιτική κτλ. Ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και οπωσδήποτε να ολοκληρωθούν και οι δεσμεύσεις ε, οι οποίες έχουν ληφθεί στις διασκέψεις κορυφής ε, σαν αυτές που μας δείχνετε προηγουμένως στις ε, διαφάνειες, διασκέψει κορυφής μεταξύ των χωρών τη Λατίνική Αμερικής, τη Καραϊβική και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι οι γνωμοδοτήσεις έχουν συγκεκριμένο ε, περιθώριο ε, μάκρους τέλο πάντων. Θα υπάρξουν όμως και τροπολογίες μέσω των οποίων οπωσδήποτε θα μεγαλώσει λίγο η γνωμοδότηση. Και εγώ δεν, έχω, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να δεχτώ τροπολογίες οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να συνάδουν με το πνεύμα της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. τον κύριο Αγουστίν. Γκερέρο. Διάφτε μέρα, συγγνώμη. ποιο άλλο θέλει το λόγο. Κάποιος συνάδελφος. Κανείς άλλος. Κύριε Διάφτε μέρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω και να ασχοληθώ με τα κεντρικότερα στοιχεία, γιατί θέλω να συσχετήσω ε, αυτά που είπε ο κύριος ε, Χουάν Μανουέλ Σαντομέ για την Ευρωσοσιάλ ε, με αυτά που είπε μόλις ο Ενρίκε. Σας συστήνω κύριε Σαντομέ να διαβάσετε την ανακοίνωση της Κομασιόν σε σχέση με τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των, των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής. Ε, είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτερες κόχες ε, μεγάλης φτώχειας βρίσκονται τελικά στις χώρες μέσου εισοδήματος ε, και η, ο διαχωρισμός των χωρών σύμφωνα με το ε, εισόδημα ε, είναι απατηλός γιατί δεν μας λέει ακριβώς τι συμβαίνει στις χώρες αυτές. Επίσης, επίσης είναι κοινό τόπος ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δείχνει χαμηλές προοπτικές ανάπτυξης για τη Λατινική Αμερική. Όσον αφορά την έλλειψη ε, ισότητας, τι ε, ανισότητε, είναι γεγονός ότι ο δείκτη ε, ένδυας και ανισορροπίας και ανισότητας έχουν βελτιωθεί σε αυτή την πλευρά του κόσμου περισσότερο από που, οπουδήποτε αλλού. Ωστόσο δεν υπάρχει γενικότερη βελτίωση της κατάστασης σε όλες τις χώρες, άρα δεν θα πρέπει ε, να σταματήσουμε την προσπάθεια. Επίσης, ε, όσον αφορά τους στόχους, ε, οπωσδήποτε ε, κεντρικός στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης, ε, η επένδυση στην καινοτομία, επίσης ε, η διαφοροποίηση των παραγωγικών δομών, γιατί είναι γεγονός διαπιστωμένο ότι τα προβλήματα είναι επίσης και απόρρια της μείωσης των ε, τιμών των πρώτων υλών. Υπάρχει επίσης και μία παράμετρος που ανέφερε ο συνάδελφος ε, Γκερέρο προηγουμένως ε, είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς που είναι ενδυμική στις χώρες αυτές. Ε, επίσης ε, η συμπερίληψη της ε, κοινωνίας των πολιτών γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στις, χώρες αυτές η κοινωνία οργανώνεται μέσω των ομάδων που πουλάνε ναρκωτικά και μέσω των μάρας, των συμμοριών. Αυτό θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Να σας πω και κάτι ανεκδοτικό αλλά μεγάλης ε, σημασίας. Εμείς ε, στην ε, ουσία ε, στην ε, Ονδούρα ας πούμε ε, εμείς θέλουμε να, να είναι υποψήφιος για το βραβείο του πρίγκιπα των Αστουριών ο, ακριβώς αυτός ο άνθρωπος στην Ονδούρα ο οποίος προσπαθεί να βγάλει τα νέα παιδιά από τα ναρκωτικά και προσπαθεί να εμφυσίσει ακριβώς αυτές τις αρχές τις ε, σωστές. Ε, επίσης να πω στον Ενρίκε ότι θα υποβάλω 7 τροπολογίες ε, τις οποίες ελπίζω να δεχτεί. Ευχαριστώ. Η Λόλα Σάντσες. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Ευχαριστούμε ε, τον ε, κύριο Σαντομέ που μας ε, είπε όλα αυτά που σχετίζονται με την εργασία του. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι αν υπάρχει μια λησμονημένη περιφέρεια και σε αυτήν την, την επιτροπή μας, αυτή είναι η Λατινική Αμερική. Το είπαμε και στους συντονιστές ότι ότι από τη στιγμή που άρχισαν να εφαρμόζονται οι αρχές της διαφοροποίησης ξεχάσαμε ε, την ε, Λατινική Αμερική και ξεχάσαμε ε, όλα αυτά που συνέβησαν την τελευταία δεκαετία στις χώρες αυτές και όπως ακριβώς έδειξαν και τα γραφήματα που μας έδειξε ο προηγούμενος ομιλητής 175 εκατομμύρια άνθρωποι στη Λατινική Αμερική ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας και αυτό από μόνο του ε, πρέπει να στρέψει την προσοχή μας εκεί. Ε, είναι γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί κάπως τα οικονομικά στοιχεία σε πολλές περιοχές ε, αλλά η φτώχεια παραμένει. Δεν θα πρέπει να δούμε τη Λατινική Αμερική μονάχα σαν ένα οικονομικό εταίρο. Θα πρέπει να δούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι. Στις μελλοντικές μας σχέσεις με την Λατινική Αμερική θα πρέπει πρέπει ε, να καταλάβουμε ότι ε, οι, ελεύθερε οι το ελεύθερο εμπόριο ε, δεν σημαίνουν αυτομάτως και καλύτερη κοινωνική κατάσταση. Αντιθέτως μπορεί να χτίσει ψηλότερα τείχη και μεγαλύτερους περιορισμούς. Επίσης εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές καταπατήσεις των ανθρωπίνων ε, ε, δικαιωμάτων σε όλες τις ε, χώρες. Ας πούμε η παράνομη κράτηση της Μιλάγρο Σάρα, η κατάσταση όσον αφορά αυτόχθονες πληθυσμούς, η ατιμορρησία εξοκολουθεί να υπάρχει. Επίσης έχουμε στην Ονδούρα την δολοφονία της Κάθερες και άλλων αγωνιστών για τα δικαιώματα των γυναικών. Επομένως, θα πρέπει να δούμε την βιώσιμη ανάπτυξη μαζί με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά την οικονομία, ε, βεβαίω εμεί συμφωνούμε γιατί ε, μέσω ε, των οικονομικών συμφωνιών τελικά το μόνο που πετυχαίνουμε όμως είναι εξαγωγική, συγγνώμη, εξορυκτική οικονομία και εξαγωγική οικονομία οικονομία. Εμείς θα θέλαμε οικονομικές σχέσεις οι οποίες θα έχουν ε, οικονομικά ωφέλη και για τις δύο πλευρές και οι οποίες ε, θα βοηθήσουν και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε ε, κοινωνικές πολιτικές μέσα από τις οικονομικές και δημοσιονομικές αρχές. Θέλουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, θέλουμε καταπολέμηση της τιμωρησία, μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, κατά καταπολέμηση της διαφθοράς, ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων ή στην κοινωνία. Επίσης θέλουμε σωστές, προοδευτικές και δικαστικές αρχές, ε, συστήματα δικαιοσύνης αμερόληπτα και δίκαια, ε, ανακατενημητικές ε, οικονομικές πολιτικές και θα καταθέσουμε λοιπόν και τροπολογίες κατά την έννοια αυτή. Επίσης, ε, για τον Χουάν Μανουέλ, ε, δύο ερωτήσεις, ε, μια και είσαι εδώ μαζί μας. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Δεκαετές είναι το πρόγραμμά σας και αφορά αρκετές χώρες, αλλά ποια είναι η άποψή σου και ποια είναι ε, ε, ε, η, θέση σου όσον αφορά τις μεγάλες προκλήσεις. Πρέπει να πω ότι η νέα εκδοχή του προγράμματος έχει ιδιαίτερη εστίαση σε θέματα φύλου. Ωστόσο θα ήθελα να μου πεις ποιες είναι οι λεπτομέρειες αυτού του σημείου καθώς επίσης και ποια είναι τα προσκόμματα τα οποία σας εμποδίζουν αποτελεσματικά να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι και η ΕΕ θα απαντούσε για το θέμα της στρατηγικής. Κύριε Φερνάντο Πόνθε, καλά το λέω. Έχετε το λόγο. Δεν, δεν έχω το όνομά σας νομίζω πολύ σωστά. Εγγραμμένο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Να σας συγχαρώ και για την εργασία την οποία ε, είδαμε σε σχέση με το πρόγραμμα Eurosocial. Θα ήθελα να κάνω και κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σας πω ότι είμαι επικεφαλής της ε, μονάδας για το Μεξικό και την ε, Καραϊβική. Εγώ βέβαια θα κάνω κάποια ε, σχόλια τα οποία αφορούν αυτέ τι χώρε για τι οποίε είμαι αλλά νομίζω ότι ισχύουν και για τη γενικότερη περιοχή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι και οι συνάδελφοί της ε, γενική διεύθυνση ΔΕΦΚΟ που ασχολούνται με την ε, συνεργασία και την ανάπτυξη μπορούν να συμβάλλουν. Όσον αφορά το Μεξικό και τι χώρε τη Καραϊβικής, τα θέματα όλα αυτά που εθίγησαν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, αναφέρθηκαν ήδη, δεν θα τα επαναλάβω. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι είναι μια στιγμή που ανοίγονται ευκαιρίες για πολλούς λόγους. Ε, ε, μεταξύ αυτών, αυτό που ε, εφημιστικά αναφέρεται αναστροφή της συγκυρίας στο Βορρά. Είναι σημαντικό λοιπόν να ενισχυθεί η διακυβέρνηση και η συμπερίληψη. Ε, ε, για τη διακυβέρνηση πολλά έχουν υποθεί αλλά και η συμπερίληψη της ε, οικονομίας και της βοήθειας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, τα ανθρώπινα δικαιώματα οπωσδήποτε βρίσκονται στο κέντρο της δράσης μας, όχι μέσα και μόνο από τις ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιβάλλουμε, αλλά και μέσα από τις καθημερινές σχέσεις με τις άλλες χώρες. Έγινε λόγος για σχέσεις μεταξύ ισοτήμων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρεσβεύουμε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντομέ να απαντήσει τις ερωτήσεις της κυρίας ε, Σάντσες. Και μετά έχω και εγώ μια ερώτηση. Ακούμε πάρα πολλά και ο Ενρίκη περισμένα πράγματα για τους ε, εργαζομένους υπέρ των δικαιωμάτων σε χώρες Λατινικής Αμερικής. Ε, για τους εργάτες στο Ζαχαροκάλαμο μου είπαν πολλές φορές ότι θίγονται από πάρα πολλές, πλήττονται από πάρα πολλές ασθένειες κλπ. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα κατά πόσο δηλαδή αντιμετωπίζετε τα θέματα αυτά στο πρόγραμμά σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το, τις γυναίκες, με τις ε, διακρίσεις λογοφύλου που ανέφερε η κυρία Σάντσες. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι ότι υπάρχει μια πατριαρχική κουλτούρα στις ε, χώρες. Είναι μια κουλτούρα ε, ανδροπρεπής, ματσίστα. Ε, και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, πολλές φορές ε, και στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί το κεντρικό πρόσκομα στη, για την προώθηση των πολιτικών που θα άρουν τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, τώρα ε, ε, είμαστε σε μια φάση όπου βλέπουμε τα αιτήματα των διαφόρων χωρών γιατί το πρόγραμμά μας προχωράει, βασίζεται στα αιτήματα που έρχονται από τις διάφορες χώρες. Έχουμε επισκεφτεί έξι χώρες και νομίζω ότι ε, όλοι, όλες λένε το ίδιο. Πρώτον θα πρέπει να ενισχυθούν ε, οι, όλες αυτές οι δομές ε, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες ε, και να τις περιβάλλουν. Είτε πρόκειται για το Υπουργείο Ισότητας, είτε πρόκειται για οργανώσεις γυναικών. Πάντως όλες αυτές οι δομές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες. Προκύπτει ότι αυτό είναι ο καλύτερο δρόμος. Δεύτερον, και αυτό είναι επίση σημαντικό, το θέμα ε, της ε, βία κατά των ε, γυναικών σε όλες τις χώρες. Φαίνεται ότι και στην Ευρώπη η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη σε ορισμένε χώρε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κοινό πρόβλημα και προσπαθούμε να βρούμε λύσει σε αυτό. Είναι θέμα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουν οι δολοφονίες γυναικών που βλέπουμε σε όλες τις χώρες της ε, Λατινικής ε, Αμερικής. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα των προϋπολογισμών δηλαδή ε, να εντάσσεται το θέμα, το ζήτημα των ε, γυναικών, η προοπτική των ε, γυναικών στους προϋπολογισμούς, να υπάρχουν ποιοτικοί δείκτες κλπ. Ναι, υπάρχουν κάποια προσκόμματα, αλλά κυρίως υπάρχουν προκλήσεις που μας οδηγούν προς τα εμπρός. Σε σχέση τώρα με τις ε, ε, φορολογικές ε, πολιτικές και τους προπολογισμούς. Νομίζω ότι το συμμερίζονται όλοι ότι έχουν υπάρξει κάποια θετικά στοιχεία και κάποιες πρόοδοι τα τελευταία χρόνια. Έχει διευρυνθεί η φορολογική βάση, όχι αρκετά η ανακατανημητική ας πούμε διάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται εδώ για μια περιοχή του κόσμου ε, όπου ε, είναι μικρότερη η φορολογική βάση και ε, είναι μικρότερη και η ανακατανομή βάση του φορολογικού συστήματος. και ε, επομένως ε, πρέπει να ε, δούμε ακριβώς την άμεση φορολόγηση. Νομίζω ότι και η ΔΕΒΚΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι και τα Ηνωμένα Έθνη και ο ΩΣΑ συμφωνούν ότι θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα της άμεσης φορολόγησης. Ένα τελευταίο και θα τελειώσω ε, η ποιότητα των δαπανών, δηλαδή θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές οι δαπάνες, πώς δαπανώνται τα δημόσια κονδύλια το δημόσιο χρήμα να πρέπει να προωθείται σε δημόσιες πολιτικές οι οποίες μπορούν να έχουν άμεσα αποτελέσματα. Ίσως μετά μπορείτε να, τα, να ολοκληρώσετε τη συζήτηση διμερώς όμως. Ε. Μάλλον θα πρέπει να συνεχίσετε διμερώς. Κοιτάζω το ρολόι μου, λέει η πρόεδρος. Κάτι πολύ γρήγορο. Δεν μου υπόθηκε πως θέλεις να μιλήσεις. Παρακαλώ πάρα πολύ γρήγορα, αν έχετε να προσθέσεις κάτι. Θα έχουμε αργότερα μια σχετική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, επίσης για το, για το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα να σας πω πως είμαστε σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένοι με το κείμενό σας και πως η συνεργασία μας ήδη υλοποιείται και πηγαίνει προς την κατεύθυνση που αναφέρεται. Για κάθε σημείο θα μπορούσα να σας δώσω παραδείγματα στα οποία εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Πολύ σύντομα και στη συνέχεια θα καταθέσω, αργότερα θα καταθέσω γραπτά σχόλια και μπορούμε να έχουμε διμερείς συνομιλίες αργότερα. Έχουμε μία σύνοδο τον Οκτώβριο. At the joint implementation as equal... Και οι μηχανισμοί βιώσιμης ανάπτυξης θα παίξουν ρόλο εκεί. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν θύλακες φτώχεια στη Λατινική Αμερική, αλλά πώς είπατε σωστά, πρέπει να κοιτάξουμε τις δημόσιες πολιτικές, το Eurosocial, όπως και πολλά άλλα προγράμματα τα οποία βοηθούν και έχουμε ένα πολύ έντονο πολιτικό διάλογο με όλες τις χώρες της περιοχής. Γι' αυτό και επιμένουμε σε μια δίκαιη και ισότιμη φορολογική και φοροεισπρακτική πολιτική ενάντια στη διαφθορά, επειδή γνωρίζουμε χωρίς αυτό. Δεν θα, είμαστε, δεν θα μπορέσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη μας να χορηγήσουν περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια στα κράτη αυτά. Πρέπει να δούμε επίσης μια προσπάθεια στις ίδιες τις χώρες να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά και να κινητοποιήσουν κονδύλια στο εσωτερικό τους. Επίσης θα ήθελα να πω πως δεν μειώσαμε τα κονδύλια μας για την περιοχή αυτή. Ανέχονται στο ίδιο ύψος με την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο. Αλλά για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική μειώσαμε τον καταμερισμό στις χώρες. Αλλά το όλο ποσό είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό δεν ισχύει για την ανθρωπιστική βοήθεια, έχετε δίκιο. Η ανθρωπιστική βοήθεια, όλος προϋπολογισμός, από ό,τι μου λένε οι συναδελφοί μας, έχει υποδιπλασιαστεί. Οπότε έχουμε, αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την ζήτηση τελευταία. Οπότε πρέπει να βελτιώσουμε την καταστασία όπου μπορούμε και μας εξηγούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια μόνο σε περιπτώσεις επίγουσας ανάγκης. Εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά με τα προγράμματα μας όπως κάνουμε στην IT όπου παίρνουμε λεφτά από την ΕΦΚΟ τα δίνουμε στους συνάδελφούς μας από την ΕΚΟ ώστε να ανταποκριθούμε σε περιπτώσεις επίγουσας ανάγκης έτσι ώστε να μπορούν τα χρήματα αυτά να επενδυθούν στην αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης με τα επιρωτικά μας προγράμματα στηρίζουμε το πρόγραμμα δράσης και για τη σύνοδο επιμένουμε να εστιάσουμε σε λίγα αλλά απτά αποτελέσματα. Μπορούμε να εργαστούμε με την περιοχή επί των ζητημάτων αυτών δεν νομίζω πως μπορώ να συνεχίσω για πολύ ακόμα, αν και θα μπορούσα να συνεχίσω να μιλώ για ώρες, αλλά ίσως μπορούμε να το κάνουμε διμερώς. Και θα λάβετε τα σχόλιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, για την επικοδομητική αυτή συμβολή. Δυστυχώς έχουμε το χρονοδιάγραμμα. Ενρίκε, έχεις τον λόγο. Δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία φορά που θα μιλήσω, αλλά θα μιλήσω σύντομα. Πριν φύγεις, πριν φύγεις, έλα παίρνω από εδώ, δεν πειράζει. Λέει στον κύριο Διευθυντεμέρα. Μέρα. Σχετικά με τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν και από αυτά που είπε και η Γενική Διευθυντεύκο. Ξέρετε, εγώ είμαι εισηγητής ε, και για την ανθρωπιστική βοήθεια και πρέπει να δούμε κατά πόσον συμφωνούμε ε, η αρχική φάση της ανθρωπιστικής βοήθειας να γίνει και φάση ανθεκτικότητας ε, ε, και αν θα ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή. Εγώ Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Αγκουστίνε και την Λόλα ε, γιατί μου είπαν ότι θα προσπαθήσουν μέσω τροπολογιών να πλουτίσουν την εκθεσή, την γνωμοδότηση. Ε, ναι, και εγώ θα σας πω κάτι που δεν είναι εύκολο να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, ε, ότι εγώ που λέγομαι ε, πλούσιος θα δεχτώ να εμπλουτιστεί η ε, έκθεσή μου. Ωραία και ελπίζω ότι έτσι κλείσαμε ωραία με αυτό το Ισπανο-Ισπανικό χειμωράκι. Ευχαριστώ. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 28 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. Με πολύ χαρά θα περιμένω να γίνει η αποστολή μας εκεί και να το ε, ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Τελευταίο σημείο για σήμερα, αλλά πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, λέει ο κύριο Σαλόμ. Α, ε, ξέχασα ε, να, σας, να ευχαριστώ τον κύριο Πρεντάβας για την βοήθεια που μου έδωσε. Ευχαριστώ ώρα των ερωτήσεων. Έχουμε τρει ερωτήσεις, έχουμε 10 με 12 λεπτά γιατί μετά πρέπει να πάμε στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΑΦΕΤ και Budget ε, για το για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Χάιντι Χάουτελα είναι η πρώτη ερώτηση. Δεν θα το διαβάσω. Ο τρόπος με τον οποίο συνεδρίασε η Επιτροπή 19 Μαρτίου για το, η Επιτροπή ΟΣΑ ε, και ΝΤΑΚ και συζήτησε τον τρόπο με τον οποίο ο ιδιωτικό τομέα θα, στην αναφέρει στην Επιτροπή ε, ΝΤΑΚ. Έχω δεν έχω τα ονόματα της, ε, των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, για την απάντηση του θέματος αυτού. Παρακαλώ, συστηθείτε. Είμαι ο Φαμπιόν Τελκρός από την ε, Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ ε, που ασχολούμαι με τα θέματα της χρηματοδότησης της ε, ανάπτυξης. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με την Ευρωβουλευτή Χάουτελα ότι τα κονδύλια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της, ε, του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης ε, και ότι θα έπρεπε να εξασφαλίζεται ότι τα κριτήρια εφαρμογής γίνονται πλήρως σεβαστά και όπως γνωρίζετε αυτά τα κριτήρια ε, έχουν επαναξεταστεί το 2015 στην Αντίσα Μπέμπα και στη Νέα Υόρκη και αυτή τη στιγμή ο ΩΣΑ ενημερώνει την ε, οδηγία για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για να, για να, να φαίνονται αυτές οι αλλαγές ε, οι συμφωνίε στην Αντίσα και στη Νέα Υόρκη δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην βιώσιμη ανάπτυξη, όπω επίση και στην ανάγκη καλύτερη χρήση τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για να αποτελέσει καταλήτη ε, τι ε, επενδύσει στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεχώ ενημερώνονται οι ορισμοί για να μπορούμε να αντικατατροπίζουμε καλύτερα το σημαντικό ρόλο των, ε, του ιδιωτικού τομέα ε, στην επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τώρα τις αρχές, ε, ο ΣΑ ε, ακολουθεί τους, τους ε, ορισμούς των υπουργών, δηλαδή ότι πρέπει ο ιδιωτικό τομέας να έχει ένα συγκεκριμένο μερίδιο, αλλά παράλληλα να, υπάρχει και μία, να υπάρχουν και κίνητρα χρήσης στις λιγότερο προηγμένες χώρες. Όσον αφορά τώρα τη μέθοδο, η μέθοδος που αυτή τη στιγμή είναι διαπραγμάτευση ε, είναι να δοθεί προτεραιότητα στην ε, προσπάθεια των δωρητών. Ε, τα μέτρα αυτά ε, για την προσμέτρηση μάλλον του υπολογισμού ε, των δωρητών, του υπολογισμού των, της συμμετοχής των δωρητών, ε, πρέπει να τα αντιπαραβάλλουμε με μέτρα αγοράς, όπως για παράδειγμα ενίσχυση της διαφάνειας και τη σημαντική ιδέα της προσθετικότητας, που σκοπό έχει να αντανακλά το γεγονός ότι οι δωρητές εφαρμόζουν αναπτυξιακή χρηματοδότηση όταν η αγορά από μόνη της δεν το κάνει. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να εγγυάται απλώς ότι οι δωρητές ε, θα καλύπτουν ε, τις ανεπάρκειες και τα κενά της αγοράς. Όσον αφορά τη χρήση των εγγυήσεων, που ήταν ένα συγκεκριμένο ερώτημα εν προκειμένου, δεν έχουμε συγκεκριμένο ποσοστό υπόψη. Ο στόχος είναι να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά των εγγυήσεων αναφέρονται δε όντως ε, στις σχετικές οδηγίες με σκοπό να δώσουν κίνητρα για τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων ε, και ένα παράδειγμα είναι η μελλοντική χρήση των εγγυήσεων ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όσον αφορά την 9η Μαρτίου και τη συγκεκριμένη επιτροπή που αναφέρθηκε η συνεδρίαση αυτή δεν κατέληξε πουθενά. Εξακολουθούν να υπάρχουν διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε να ολοκληρώσει εργασίε της το δυνατόν. Η κυρία Χάουτελα, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αυτή. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην, στον ΟΣΑ ε, θα μπορέσει να υπερασπιστεί μια γραμμή που υπερασπίζεται την ακαιρεότητα και την αξιοπιστία της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά έχουμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα όσον αφορά το ερώτημα των κρυμμένων επιδοτήσεων όσον αφορά τις εγγυήσει εξαγωγών και έχω παρατηρήσει ότι φαίνεται να υπάρχει μία ε, ανισορροπία μεταξύ ε, τη, των ε, ε, ε, οργανώσεων, ανα, των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης και της, των, μέσων επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. μήπως μπορείτε να μας πείτε περισσότερα από αυτού. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο επίπεδα ε, πρέπει να ε, σε δύο επίπεδα πρέπει να αναφερθώ για να απαντήσω. Το πρώτο επίπεδο είναι γενικό, ότι φυσικά θα ισχύουν τα κριτήρια όσα ε, για τα, τα κριτήρια συγγνώμη, της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα δικαιούχος πρέπει να αναφέρεται ως χώρα δικαιούχος της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Οπότε τότε η εξαγωγική πίστοση θα έπρεπε να περνάει από, μια, από έναν επίσημο οργανισμό. Το ερώτημα τώρα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή ε, αυτή η πίστοση ε, θα ε, είναι όντως μια εξαγωγική πίστοση και όχι μια κρυμμένη επιδότηση. Δύο μεταβλητές ακόμη διαπραγματευόμαστε. Το πρώτο είναι το επιτόκιο που θα προσφέρετε και το δεύτερο η το επίπεδο ποσοστού έκπτωσης που θα εφαρμόζεται στο, στο μέσο. Ε, και εμείς είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι οποιαδήποτε, οποιοδήποτε κέρδος ε, υπάρξει ε, θα πρέπει να πληρωθεί ως αρνητική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια να επιστραφεί ε, στις χώρες με αποτέλεσμα να είναι απολύτως ουδέτερη η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο ερώτημα. Από τον Ενρίκη Γκερέρο Σαλόμ για την πείνα στην Ιγυρία, το, South, το, κάτω, το, συγγνώμη, Νότιο Σουδάν, την Αιθιοπία, τη Σομαλία και την Ιεμένη. Ε, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο περισσότερα για το τι προγραμματίζεται. Η κυρία Μαγιό είναι εδώ για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όπως είπε και ο Επίτροπος την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να ανησυχεί έντονα για την ανθρωπιστική κατάσταση στην λίμνη του Τσάτ και ιδίω στην Γυρία, όπου πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τέλος του 2015 ήδη προειδοποίησε για λοιμό αλλά η προειδοποίηση αυτή δυστυχώς δεν ελήφθη σοβαρά και δεν υπήρξε επαρκής διεθνής κινητοποίηση και συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε σταδιακά από το 2014 την υποστήριξή της προς την περιοχή της λίμνης του Τσάτ και την Ιγυρία, δίνοντας υποστήριξη διάσωσης και διατροφής και προστασίας της υγείας πέρυσι 62 εκατομμύρια ευρώ επιμερίστηκαν στην Ιγυρία για δραστηριότητες αυτού του είδους που αποτελούν μέρος της στρατηγικής μας για το 2017 επίσης. Ο αρχικός καταμερισμός μας για την κρίση της δήμης του Τσάντ ήταν 55 εκατομμύρια και ζητήσαμε άλλα 55 εκατομμύρια, άλλα 50 συγγνώμη, από το αποθεματικό επίκουσας ανάγκης για να συνεχίσουμε να δίνουμε βοήθεια και να επιτύχουμε μια από κοινού προσέγγιση με τους εταίρους μας, ιδίως στην βόρειο-ανατολική Νιγηρία, όπου συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας της αναπτυξιακής βοήθειας, το λεγόμενο πακέτο αμπόρνου, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού αλλά και του δημόσιου τομέα στην περιοχή. Το πρόγραμμα αποσκοπεί να αποτελέσει επίδειξη του, της ύπαρξης του συνδέσμου μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης. Το είδαμε στον Πόρνο Ακουατάι. Θα έχει διάρκεια 48 μηνών και πέρα από την επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται ακόμα περιλαμβάνει υποστήριξη για την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών κυρίως στην περιοχή, στον τομέα της υγείας, της παιδείας και της διατροφής σε το, περιοχές μετεγκατάστασης ή όπου έχουμε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες. Αποσκοπεί επίσης τη δημιουργία και παροχή υποστήριξης για την διαβίωση, δυνατότητες απασχόλησης και δημιουργίας κοινωνικής προστασίας και αυτή η υποστήριξη αποσκοπεί κυρίως σε νέους και γυναίκες. Και τέλος, ο στόχος είναι επίσης η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης υπό την έννοια της αύξησης βιώσιμων δημόσιων υπηρεσιών όσον αφορά τις βασικές υπηρεσίες. Όσον αφορά το Νότιο Σουδάν, επί του παρόντος 82 εκατομμύρια καταμεριστήκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για επιχειρήσεις βοήθειας 42 εκατομμύρια εκ των οποίων καταμερίστηκαν τον Δεκέμβριο για την αντιμετώπιση κυρίως της επιστηστικής κρίσης περιλάμβανε επίσης την παροχή επίγουσας επιστηστικής βοήθειας σε πληθυσμούς που ζουν σε περιοχές όπου όντως στις 20 Φεβρουαρίου εντοπιστήκε φαινόμενα λοιμού. Άλλα 100 εκατομμύρια από το EDF ανακοινώθηκαν από την Επίτροπο Μογκερίνη και από τον Επίτροπο Στυλιανίδη για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης λόγω της σύραξης στο Νότιο Σουδάν. Από τα χρήματα αυτά 30 εκατομμύρια θα απευθυνθούν στη διάσωση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων στο νότιο Σουδάν. Θα παρασκευθεί βοήθεια, παραδείγματο χάρη, για την προστασία γυναικών και παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο και για την αντιμετώπιση φαινομένων οξίας, προβλημάτων διατροφής θα χρησιμοποιηθούν επίσης χρήματα για την υποστήριξη στις γειτονικέ χώρες, την Αιθιοπία, την Ουγάντα, την Κένια και το Σουδάν, για να παρασκευθεί συνεχής βοήθεια για την αντιμετώπιση των αναγκών των Σουδανέζων προσφύγων, των νότιο Σουδανέζων προσφύγων, συγγνώμη, που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις αιστείες τους. Όσον αφορά τη Σομαλία, 65 εκατομμύρια ευρώ ζητήθηκαν από το αποθυματικό επίγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που προκλήθηκε από την ξηρασία στην Σομαλία, το Σουδάν και την Κένια, εκ των οποίων 45 εκατομμύρια ευρώ θα ξοδευτούν για την υποστήριξη διάσωσης του πιο ευάλωτου πληθυσμού στη Σομαδία, όπου ήδη έχουμε έναν συναγερμό πρόλημου. Βασικές προτεραιότητες είναι η επίγουσα επιστηστική βοήθεια και αντιμετώπιση της κακοδιατροφής, του υποσυντισμού, συγγνώμη, επίσης και υποστηρίξη για το πόσιμο νερό, Επίσης όσον αφορά τα μέσα έχουμε δια... εμβάσματα χρημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την τόνωση των τοπικών οικονομιών έτσι ώστε οι πληγόμενοι πληθυσμοί να έχουν περισσότερες επιλογές. Επίσης, σε όλες τις προσπάθειες αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει, καταβάλει ξεκαθαρές προσπάθειες για καλό συντονισμό μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο τα άμεσα αποτελέσματα αλλά επίσης τα αίτια του υποσυντισμού όσον αφορά την Ιεμένη. Η παροχή βοήθεια στην Ιεμένη είναι μια κούρσα ενάντια στον χρόνο. Θα έχετε ενημερωθεί από την Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών που τόνισε ότι το 70% του πληθυσμού είναι 18,2 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται άμεσα βοήθεια και 7 εκατομμύρια δεν γνωρίζουν πώς να αποκτήσουν πρόσβαση στο επόμενο γεύμα τους παρά το γεγονός πως η Γεμένη αποτελεί τη μεγαλύτερη διατροφική κρίση αυτή τη στιγμή, κρίση αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έχουμε μια, στις 24 Απριλίου μια σύνοδο στην Γενέβη, την οποία, στην οποία συγκαλεί η Ελβετία και η Σουηδία. Από την έναρξη της σύραξης η Επιτροπή κινητοποίησε 120 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση της κρίσης της Το ίμιση του προϋπολογισμού αυτού χρησιμοποιήθηκε για την επιστηστική βοήθεια και το άλλο ίμιση για τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε ίδρευση για υγιεινή και για την υποστήριξη για βασική στέγη. Η υποστήριξη κατά προτεραιότητα απευθύνεται σε περιοχές όπου ο πληθυσμός είναι πιο ευάλωτος όπου τα επίπεδα του σοβαρού υποσυτισμού είναι τα πλέον υψηλά. Καθώς η σύραξη δεν περιορίζεται πλέον σε συγκεκριμένες περιοχές και τα μέτωπα αλλάζουν συνέχεια, η απόκρουση εστιάζει σε περιοχές επίγουσες ανάγκης και είναι ευέλικτη γεωγραφικά κινητοποίησή του αποθεματικού αν βοήθειας για την Ιεμένη θα συμβάλλει στη συνέχιση της υποστήριξης έτσι ώστε να συνεχίσει να χρηματοδοτείται να συνεχιματοδοτούν να θέσει χρήσιμες ε, δραστηριότητες στην περιοχή. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, λέει ο κύριο Γκερέρε. Ήταν εξαντλητική η πληροφόρηση. Θα ήθελα γι' αυτό να ευχαριστήσω την Κομισιόν. Και να καλωσορίσω και τον Ζαχαρία που τον ξέρω. Εγώ ακριβώς υπέβαλα την ερώτηση αυτή έτσι ώστε να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε ε, στην αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος της, ε, του λοιμού που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες. Κάτι ακόμη για την κρίση αυτή, τα διδάγματα που μπορούμε να τλήσουμε. Εγώ ενημερώθηκα για το θέμα αυτό ε, για τον ενδεχόμενο ενός ε, λοιμού το περασμένο καλοκαίρι, λίγο πριν το καλοκαίρι. Το Δεκέμβριο του 2015 υπήρχαν ε, προειδοποιήσεις ότι θα υπήρχε εξηρασία και ότι ο κόσμος ήταν ευάλωτος αυτό που με ρωτάνε εμένα οι ψηφοφόροι μου είναι για ποιο λόγο δεν κάναμε τίποτε, ε, γιατί δεν ήμασταν προετοιμασμένοι ενώ το, το ξέραμε ότι ερχόταν. Γιατί δεν είχαμε έτοιμους κάποιους μηχανισμούς να αντιμετωπίσουμε. Ίσως δεν πρέπει να το θέσουμε αυτό σήμερα, αλλά σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή είναι το ερώτημα που πρέπει να τεθεί. Γιατί σε κάποιες χώρες, ας πούμε στην Αιθιοπία, ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι από τις άλλες χώρες ε, Εντάξει, για μένα είναι εντελώ διαφορετική περίπτωση. Είναι εμπόλεμη ζώνη, το Σουδάν επίση, αλλά ε, το φαινόμενο Ελνίνιο και οι, κλιματικοί, οι κλιματικέ συνέπειε μήπω επηρεάζουν, ε, ίσω πρέπει και ε, με τον Επίτροπο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πώ μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό. Γιατί πραγματικά μα πάει πίσω σε μια εποχή στην οποία θεωρούσαμε ότι έπρεπε να έχουμε ξεπεράσει όσον αφορά την Αφρική. Ωραία, μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και με τον Επίτροπο Στυλιανίδη και να ακούσουμε περισσότερα για το ε, πώς δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Να μάθουμε το μάθημά μας γιατί είναι μια πραγματικά πολύ θλιβερή κατάσταση. Τελευταίο ερώτημα είναι για την εξάλληψη της πολιομιελίτιδας. Ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό ε, έχουμε κάποιες ε, γραμμές προπολογισμού, ειδικότερα για τις χώρες στι οποίε εξακολουθεί να υπάρχει ομιελίτιδα, ε, Νιγηρία, Πακιστάν, Αφγανιστάν. Και ρωτάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα γίνει. Γιατί υπάρχει νομίζω η ελπίδα ότι μπορούμε να την εξαλείψουμε. Υπάρχει αυτή η ελπίδα τώρα. Ιαν Παλιέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι επικεφαλή ε, τη ομάδα για την υγεία τη Γενική Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ. Θα ήθελα να πω ότι εμεί παραμένουμε απολύτω δεσμευμένοι για την εξάλληψη τη πολιομιελίτιδα. Ξέρουμε ότι εξακολουθεί να εφίσταται σε περιοχέ, όπου ε, δεν είναι πάρα πολύ καλά, ε, είναι εντελώς αποτυχημένα τα συστήματα τακτικής, τακτικού εμβολιασμού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 στις 17 χώρες ε, στις οποίες έχουμε επικεντρωθεί ε, συμπεριλαμβάνονται η Νιγηρία, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Είναι οι δύο περιοχές, ε, η Βόρεια Νιγηρία και η μεθοριακή περιοχή ορεινή μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Εκεί εξακολουθεί να εφίσταται η πολιομιελίτιδα. Όσον αφορά την Νιγηρία, το Φεβρουάριο αποφασίσαμε επιπλέον 20 εκατομμύρια να εκταμιεύσουμε για την προσπάθεια ελέγχου της πολιομήλικης μέσω του διμερούς ενδεικτικού προγράμματος αυτού του δημοσιονομικού πολιετούς πλαισίου και έχει να, αυτό ε, συνδυάζεται με την πρωτοβουλία για την εξάλληψη της ε, πολιομιλίτιδας και της προσπάθειας μετάβασης της ε, χώρας σε έναν κόσμο χωρίς πολιομιλίτιδα. Για παράδειγμα, η Κάποιοι έχουμε διαθέσει και ανθρώπινους πόρους για την προσπάθεια αυτή. Ε, στο Αφγανιστάν εδώ και πολλά χρόνια έχουμε ε, εντοπίσει αυτό το πρόβλημα. Από το 2016 ε, μέχρι το 2020 έχουμε πει γύρω στα 277 εκατομμύρια να διατεθούν για την προσπάθεια αυτή, κυρίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών με σκοπό την εξάλληψη, την εξάλληψη της πολιομιελίτιδας. Έχει ήδη ένα σύστημα το Αφγανιστάν πλέον υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας ε, για την ε, επέκταση του προγράμματος εμβολιασμού με ε, βασικό στόχο την πολιομιελίτιδα Επίσης, ε, να σας πω ότι δεν υπάρχει προχρηματοδότηση για την ώρα για το θέμα αυτό στο τρέχον, πολιο, στο τρέχον δημοσιονομικό, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όμως στην ενδιάμεση αναθεώρηση μπορεί να το λάβουμε αυτό υπόψη και αν υπάρχει ανάγκη να ε, διατεθούν κάποια ποσά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για, αυτήν, ε, την, για αυτές τις παρατηρήσεις. Περνάμε τώρα στο σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης που είναι τα διάφορα. Δεν βλέπω κανένα να θέλει να θέσει τίποτε από τα διάφορα. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι θα κλείσω την επίσημη μας συνεδρίαση γιατί θα πάμε στην, Επιτροπή, της Επιτροπής στην συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών για να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 24 Απριλίου επόμενη συνεδρίασή μας, 3 η ώρα το μεσημέρι, στις Βρυξέλλες. Αυτά. Κυρίσω λοιπόν το πέρα στη συνεδρία. ευχαριστώ τους διερμηνείς ε, και σας υπενθυμίζω ότι πάμε τώρα στο 2Q2, στο άλλο κτίριο, για ε, την συνεδρίασή μας με την Επιτροπή Εξωτερικών. Ευχαριστώ.